Αγαπητοί συνάδελφοι, πάρτε θέσεις. Θα ξεκινήσουμε με τις ψηφοφορίες. Έχουμε αργήσει. Έξι λεπτά αργήσαμε. Γρήγορα. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι σημερινή συνεδρίαση την πρωινή. Σωστά διαπιστώσατε πως η νομοθετική μας δουλειά δεν καταλαμβάνει την πλειοψηφία του χρόνου. Αλλά, αλλά δεν φταίνει οι βουλευτές. So, das ist aber nicht unbedingt αλλά αυτό δεν οφείλεται στους ε, βουλευτές αλλά στο έργο της ε, Κομισιόν που πρέπει να έχει και αντίδραση ε, και από εμάς. Βεβαίως Όλα αυτά οδηγούν δικαίως σε συζήτηση επί κάποιων θεμάτων. Αλλά θα ήθελα να σας παρακαλέσω να αλλάξει. Θα ήθελα να σας πω το εξής. Για επίμαχα θέματα υπάρχει και η δεύτερη ανάγνωση που μπορούμε να δούμε τα θέματα με μεγαλύτερη ε, λεπτομέρεια. Και δεν είναι και δημοκρατική διαδικασία κατά την άποψή μου η συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Ευχαριστώ. Χόρστ Σνέλχαρτ η τακτική κοινοβουλευτική διαδικασία νομίζω καθιστά πιο ορατή την Επιτροπή μας από μια συμφωνία στην πρώτη ανάγνωση. Και παρακαλώ, τα συζητήσαμε με τους ε, συντονιστές, απευθυνθείτε στον συντονιστή της εμπιστοσύνης σας για να ε, συζητήσετε το έργο της Επιτροπής. Αλλά το είδαμε, 25% του χρόνου μας είναι νομοθετική εργασία. Πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το πράγμα και θα το δούμε στην συνεδρίαση των ε, συντονιστών. Έχω άλλη μία... Α, ε, άλλο ένα συνάδελφο, τον κύριο Ταταρέλα που θέλει να παρέμβει. Mike θα, ήθελα να ψηφίσουμε πρώτα το δικό μου θέμα. Γιατί έχω να ψηφίσω και σε άλλη αντιπροσωπεία. Πρόταση, είναι σύντομη η έκθεση. Δεν δουλεύει η διερμηνία προς τα δανέζικα. Σουηδικά εντάξει, Ισπανικά δεν είχατε, μάλιστα. Προτείνω να το δούμε δεύτερο θέμα. Δύο ανακοινώσεις ακόμα έχω να κάνω ε, πλην της ε, ψηφοφορίας. Έχουμε τους αντιπροέδρους εδώ πέρα, τους ε, συναδέλφους, από τους οποίους είναι μεγάλη τιμή για εμάς πως κάποιος θα γίνει πρόεδρος κράτους, ο συνάλφος Γιάννος Άντερ, ο οποίος προτάθηκε στις 17 Απριλίου και στις 2 Μαΐου θα εκλεγεί, από ό,τι φαίνεται, και εύχομαι στον συνάδελφο καλή δύναμη για τα νέα του καθήκοντα. Η καιρή είναι δύσκολη και του το είπα βεβαίως ε, και σε μια προσωπική συζήτηση και έχουμε συνεργαστεί από κοινού και θα τολμήσω να πω κάτι στα Ουγγρικά. Καλή επιτυχία κύριε Πρόεδρε. Καλή επιτυχία στο νέο σας αξίωμα. Έχετε το λόγο. Ε, ευχαριστώ. Θα ήθελα και εγώ να σας πω ευχαριστώ πολύ στα γερμανικά, κύριε Πρόεδρε. Και να ευχαριστήσω όλα τα μέλη της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ τον κύριο Γιώ τον προηγούμενο πρόεδρο Ήμουν 19 ε, χρόνια πολιτικός στην ε, χώρα μου, το 1990 μέχρι το 2009 και τα τελευταία χρόνια δούλεψα και εδώ τρία χρόνια ε, και αυτά τα τρία χρόνια ήταν και μου δώσανε πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία για, για κάποια θέματα τα οποία δεν τα είχα διεξέλθει στην προηγούμενη μου σταδιοδρομία. Ε, είμαι νομικός και είχα εξειδικευθεί σε θέματα δημοσίου δικαίου στη χώρα μου, οπότε ε, η δική σας επιτροπή βέβαια έχει τεράστιο φάσμα θεμάτων, υγεία, υγιεινή, ε, ασφάλεια, περιβάλλον, τόσο τόσα πολλά θέματα. Οπότε νομίζω ότι και αυτό παρουσιάζει πάρα πολύ ενδιαφέρον και εμπλουτίζει την εμπειρία μου. Τρεις εκθέσεις μου ανετέθησαν ε, όσο ε, δούλεψα εδώ και αυτές ήταν πολύτιμες, έμαθα πάρα πολλά, σας ευχαριστώ όλους. Κάθε φορά με μάθαιναν πολλά πράγματα και με βοηθούσαν οι σκιώδες εισηγητές ε, σε αυτή τη διαδρομή των τριών ετών και είμαι σίγουρος ότι θα συνεχθούμε στο μέλλον ξανά κάπου αλλού και θα έχουμε να πούμε πολλές ιστορίες από το παρελθόν και βεβαίως το Ρίο θα τα ξαναπούμε σε δύο μήνες γιατί εκεί θα εκπροσωπήσω τη χώρα μου. Ελπίζω εκεί να δω όσο γίνεται περισσότερους συναδέλφους από σας Σας ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε την ευκαιρία να έρθω. και χίλια συγγνώμη που θα μείνω για τι εφορίε, γιατί έχω, έχω υποχρεώσεις και πρέπει να φύγω. Ευχαριστώ. Ένα συνάδελφος ε, ζήτησε τον λόγο, ο Ρίχαρτ Τζέμπερ, συντονιστής του ΕΛΚ. Έχετε τον λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, χωρίς να μακρηγορήσω, νομίζω πως ε, δεν είναι κάθε μέρα που ε, ένας συνάδελφός μας γίνεται πρόεδρος χώρας Θέλω λοιπόν να ευχαριστήσω τον Ιάννους για την εξαιρετική του εργασία και εξ ονόματος του Πέτερ Λίζε. Ήδη με προσέγγισαν και έδωσα και εγώ συνεντεύξεις για το έργο του Γιάννου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Δύο ερωτήματα ετέθησαν. Πρώτα απ' όλα γιατί εργάστηκε στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και δεύτερον εάν θα είναι ικανός να επιβληθεί του Όρμπαν. Για το πρώτο ερώτημα ε, είπα πως είναι ένας εξαιρετικός νομικός αλλά αν θέλει κάποιος ε, να κάνει κάτι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να πάει στην νομοθετική επιτροπή και η Επιτροπή Περιβάλλοντος είναι η νομοθετική επιτροπή από εδώ πέρα περνάει περισσότερη νομοθεσία και άρα ο Γιάννος ε, θεωρώ πως έκανε τη δουλειά του εξαιρετικά και αποτελεσματικά. Για το δεύτερο ερώτημα, αν θα καταφέρει να επιβληθεί του Όρμπαν, είπα πως κατάφερε σε πάρα πολύ σύντομο καιρό όσον αφορά το Σεβέζο 3 να επιτύχει πολιτικό συμβασμό και εδώ μέσα και με το Συμβούλιο που δείχνει τη διαπραγματευτική του ικανότητα, την ικανότητα συμβιβασμού και θεωρώ πως ως πρόεδρος θα ωφελήσει την Ουγγαρία γιατί υπάρχουν αυτή τη στιγμή κάποιες εντάσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι θετικό να υπάρχει στην κορυφή της χώρας κάποιος άνθρωπος που ξέρει πώς δουλεύουμε εδώ μέσα, που ξέρει πώς σημαντική είναι η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση, που ξέρει πώς σημαντικό είναι να τηρούνται οι ευρωπαϊκοί κανόνες αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Γι' αυτό χαίρομαι πάρα πολύ για το ότι θα ε, καταλάβει σε λίγο αυτό το αξίωμα. Θα ήθελα λοιπόν να προκαλέσω τον πρόεδρο προσεχώς όταν θα υπογραφεί η έκθεση σε Βέζο 3 να έρθει να την υπογράψει. Δεν νομίζω πως θα ήταν άσχημο. Σε ευχαριστούμε λοιπόν ακόμη μια φορά Γιάννος και εύχομαι και σε σένα και στην Ουγγαρία κάθε επιτυχία για το μέλλον. Ευχαριστώ, Ρίχαρτ Σέμπερ. Πολύ καλή αυτή η πρόταση και δεν νομίζω να έχει κανείς αντίρρηση, οπότε αποφασίστηκε. Κύριε Πρόεδρε, καλή επιτυχία σας εύχομαι στα νέα σας καθήκοντα και καλή τύχη. Ja, der Ένας φεύγει, ένας έρχεται. Είχα καλωσορίσει το πρωί την συνάδελφο από την Κροατία, την, από τη Σοσιαλδημοκράτη, τη Ρωμάνα Γιάκοβικ. Διευρύνεται το ευρωπαϊκό μας ε, σπίτι. Καλώς ήρθατε λοιπόν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και καλώς ήρθατε στην μεγαλύτερη νομοθετική επιτροπή, καλά τα λέει ο Ρίχαρτ τη σημαντικότερη νομοθετική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Καλή αρχή σας, εύχομαι και καλή συνεργασία με όλους μας. Καλώς ήρθατε. Οπότε τώρα περνάμε στην ημερήσια διάταξη ξανά, ψηφοφορίες, έχετε όλοι τις κάρτες σας. Ξεκινάμε με το πολιετέ σχέδιο για το απόθεμα Σολομού της Βαλτικής και την αλλιευτική εκμετάλλευση αυτού. Και περνάμε στην πρώτη συμβιβαστική τροπολογία, την παριθμόν 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Περνάμε στην τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Μετά περνάμε στην υπαρχμόν 30 υπέρ κατά αποχές δεκτή. 31 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 33 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 32 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 6 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Να επαληθεύσουμε. Να επαληθεύσουμε την παρθμόν 6. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Δεκτή με 37 ψήφου, υπέρ. 34 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 35 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 36 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 40 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 41 υπέρ κατά αποχές Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Να το επαληθεύσουμε ηλεκτρονικός. 43. 43 ψήφισμα. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 30 υπέρ και κατά απορρίπτεται. 44 υπέρ. Κατά. Εποχές απορρίπτεται. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται να επαληθεύσουμε την υπαριθμόν 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Υπάρχει κάποιος παραπάνω από τους σοσιαλδημοκράτες. Τώρα είναι εντάξει. 31 υπέρ, 30 κατά. Οπότε καλά κάναμε και το επαληθεύσαμε. Περνάμε στη 45. Όχι. Μόνο το δεύτερο μέρος της 45. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Περνάμε. Στην 46. Ποιος είναι υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεν είναι σίγουρο ενδιαφέρουσα πάντως ψηφοφορία να επαληθεύσουμε λοιπόν την 11 Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ, 29 κατά. Δεκτή. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 12 υπέρ κατά αποχές δεκτή και περνάμε στην 50 ως προσθήκη υπέρ κατά αποχές δεκτή προφορική τροπολογία του εισηγητή Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Θα ξαναρωτήσω. Ποιος είναι υπέρ της προφορικής τροπολογίας. Παρακαλώ, σηκώστε το χέρι. Κατά. Αποχές δεκτή. 50, όχι 53. 53 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 53 ψήφισαν όλοι πέρας 53 την 53 ψηφίζουμε ...37 υπέρ 23 κατά ψηφίζουμε τώρα, όχι 54 καταπίπτει. Και περνάμε σε άλλη μια προφορική τροπολογία του εισηγητού. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Μετά περνάμε στην 57 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 59 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 60 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 61 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 63 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 υπέρ κατά αποχές δεκτή 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και περνάμε σε μια προφορική τροπολογία την υπαριθμόν 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές ε, νομίζω ότι πέρασε, αλλά θα την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 37 υπέρ, 22 κατά. Εγκρίνεται. Παραρτήματα. 68 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ κατά αποχές δεκτή ε, διολογικές σκέψεις 23 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές δεκτή Ένα υπέρ κατά αποχές δεκτή Δύο υπέρ κατά αποχές δεν είμαι σίγουρος να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά έρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 36 υπέρ 23 κατά. Παρεμβαίνει ο Καρλ Σλούτερ, ήταν σαφές, αλλά δεν φαινόταν από εδώ πάνω. Mhm. Dann kommen wir auf drei. Mhm. Okay, 26. Νούμερο 3. Τρία. Παριθμόν 3. Υπέρ. Κατά αποχέ δεκτή. 27 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Καταπίπτει. 29 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή και περνάμε στην τελευταία ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά ψήφισαν όλοι πέρας 56 υπέρ 6 κατά καμία αποχή συγχαρητήρια στον Καρλ Σλούτερ. So, jetzt geht's weiter. συνεχίζουμε με την έκθεση τα παρέλια. Λοιπόν, έχουμε ε, σκάφη αναψυχής και κινητήρες θαλάσσι. Ξεκινάμε με τροπολογία 6. Υπέρ, κατά. Απορρίπτεται. Δεν ήταν σαφές νομίζω το τι πράγμα ψηφίζουμε. Ψηφίζουμε το σημείο 14 της ημερήσιας διάταξης. Το φέραμε μπροστά γιατί ο κύριος Ταταρέλα πρέπει να πάει σε άλλη επιτροπή. Και επειδή δεν υπάρχουν πολλές αντιρρήσεις, το 14 έρχεται πιο μπροστά. Και ψηφίζουμε τώρα το σημείο, την τροπολογία 6, πρώτο. Α, ποιος είναι υπέρ λοιπόν. Κατά. Όχι. Αποχές απορρίπτεται. Περνάμε στο 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 8 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 9 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 11 υπέρ κατά αποχές θα επανεξεταστεί. Να την ξαναδούμε λοιπόν την 11 η άρχη ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 24 υπέρ 37 κατά απορρίπτεται. Περνάμε λοιπόν Okay. Dann geht's weiter. Στην 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 14 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή τελική ψηφοφορία άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 56 ε, υπέρ κανείς κατά συγχαρητήρια κύριε Ταταρέλα Dann kommen wir jetzt wieder zum Tagesordnungspunkt Περνάμε ξανά στο 10. Ελαττωματικά εμφυτεύματα στήθους από γέλη σιλικόνης παρασκευόμενα από την ε, παρασκευαζόμενα από τη γαλλική εταιρεία PIP. Περνάμε κατευθείαν στην ψηφοφορία. Είναι όλοι έτοιμοι. Ξεκινάμε με την 26 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή 27 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 28 υπέρ κατά αποχές δεκτή 29 υπέρ κατά αποχές δεκτή 30 χωριστή ψηφοφορία μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 31 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές να ξαναψηφίσουμε παρακαλώ την 33 υπέρ κατά αποχές νομίζω με ισχυρή πλειοψηφία εγκρίνεται Α, να επαληθεύσουμε άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε 38 υπέρ 23 κατά δεν φαινόταν από εδώ. Παρακαλώ λοιπόν να σηκώνετε ψηλά το χεράκι. Υπέρ κατά η αποχή. Περνάμε στην 34 σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Περνάμε στην 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 38 υπέρ κατά αποχές Τι; 40 σε δύο μέρη και ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο μέρος υπέρ κατά αποχές δεκτή 41 υπέρ κατά αποχές δεκτή 42 υπέρ κατά αποχές δεκτή 43 υπέρ κατά αποχές Να επαληθεύσουμε την 43 ηλεκτρονικά. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 39 είπε. Υπέρ 23 κατά, οπότε γίνεται δεκτή. Ζιλ Πανιό κατόπιν 44 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβιβαστική 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή οπότε περνάμε στην 51 υπέρ κατά αποχές δεκτή 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται περνάμε μετά στην 53 υπέρ κατά αποχές εκτί 54 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 56 55 θέλετε να την ψηφίσουμε ηλεκτρονικά μάλιστα Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 30 υπέρ, 30 κατά. Απορρίπτεται. Ε, φαινόταν. 56 υπέρ κατά αποχές δεκτή να επαληθεύσουμε. Να επαληθεύσουμε. Την 96 Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 32 υπέρ. 29 κατά. Καταπίπτει λοιπόν η 57 και συνεχίζουμε με την 58 υπέρ κατά αποχές δεκτή 59 υπέρ κατά αποχές να το ξαναδούμε ηλεκτρονικά την 59 ε, ψήφισαν όλοι Πέρας. 35 υπέρ, 27 κατά, δεκτή. 60 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 61 υπέρ, κατά, αποχές δεκτή. 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται και μετά περνάμε στην 63 με προφορική τροπολογία ποιος είναι υπέρ με την προφορική τροπολογία κατά αποχές δεκτή 64 υπέρ κατά αποχές δεκτή 65 υπέρ κατά αποχές δεκτή 66 είναι γλωσσική υφής υπέρ κατά αποχές δεκτή 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 67 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 68 υπέρ κατά Αποχές απορρίπτεται 71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 70 γλωσσική υπέρ κατά αποχές δεκτή 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 73 υπέρ κατά αποχές δεκτή 74 υπέρ κατά αποχές δεκτή 76 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 77 υπέρ κατά αποχές δεκτή 78 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 79 υπέρ κατά αποχές δεκτή 80 υπέρ κατά αποχές δεκτή 81 υπέρ κατά αποχές δεκτή 82 υπέρ κατά αποχές δεκτή 83 υπέρ κατά αποχές δεκτή και περνάμε στα εκτιμώντας Τροπολογία 1 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 2 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 3 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Υπέρ, 4 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 5 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 10 υπέρ κατά αποχές δεκτή 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 υπέρ κατά εποχές απορρίπτεται 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 17 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτό μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ψηφίζουμε κατόπιν την 19 υπέρ κατά αποχές δεκτή 20 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε την 20 ηλεκτρονικά 20 elektronisch, haben alle abgestimmt. Abstimmung ist... 20, πέρας της ε, ψηφοφορίας. 15 υπέρ, 45 κατά. Σηκώνετε το χεράκι την άλλη φορά για να βλέπει και ο πρόεδρος. Για να μην το επαληθεύουμε. 21 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ε, ξεκάθαρα. 22 ε, υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 24 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 25 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε την 25. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 31 υπέρ. 28 κατά. Και περνάμε στην τελική ψηφοφορία, ηλεκτρονική. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 62 υπέρ, κανένας κατά, Αμία αποχή. Συγχαρητήρια στον ε, συντάκτη, καλή δουλειά. Νομίζω θα πάει μια χαρά στην Ολομέλεια. Συνεχίζουμε. Jetzt geht's weiter mit dem Tagesordnungspunkt 11. 11 γεωγραφικέ ενδείξεις αρωματισμένων αμπελοϊνικών προϊόντων. Και περνάμε στην ε, ψηφοφορία για, Τροπολογία 3 υπέρ. Υπέρ. Κατά. Κατά. Άποχες. Εγκρίνεται. 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 17 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 7 υπέρ όχι όχι, συγγνώμη. Άγκρι 5. Άγκρι 5 πρώτα. Πρώτα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Και τώρα η 7. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 8. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 18. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 19. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ε, ελέγχουμε τη 19. Ε, ελέγχουμε ηλεκτρονικά. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέραση της ψηφοφορίας. 32 υπέρ, 27 κατά. Γίνεται δεκτή 19. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 9. Άγκρι 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Άγκρι 20. Υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. 21. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Άγκρι 10. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 22. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 24. Υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. Πάμε στην 25. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26 υπέρ, κατά, αποχές, Απορρίπτεται. 27, 28, 29 και άγκρι 11. Όλοι, όλες οι ίδιες είναι. Ψηφίζουμε υπέρ, κατά, άποχες, δεκτές. 30 υπέρ, κατά, άποχες, δεκτή. 32 υπέρ, κατά, άποχες απορρίπτεται 33 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 35 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 36 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 37 38 άγκρι 12 ίδιες είναι ψηφίσουμε μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται 39 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 40 υπέρ κατά άποχες δεκτή. 41 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 42 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 43 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 44 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται 46 υπέρ κατά αποχές δεκτή 47 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 49 υπέρ κατά δεκτή 50 υπέρ κατά αποχές δεκτή άγκρι 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή άρτηρη 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 51 Καταπίπτη. 52 υπέρ κατά αποχές δεκτή 53 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 13. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 55. Ξεχωρίστα τμήματα. Ναι, ναι, ναι. Ψηφίζουμε μόνο το δεύτερο τμήμα. Δεύτερο τμήμα του 55. Ψηφίζουμε υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 56 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Άγκρι 17 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 14 υπέρ. Κατά. Έγινε λάθος. Πρέπει να ψηφίσουμε την άγκρη 18. Ποιο είναι υπέρ του άγκρη 18. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Και τώρα ψηφίσουμε το 14. Λέει ο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 15 και 16 μαζί ψηφίζουμε υπέρ, κατά, αποχές, δεκτές. 58 αγρι 20 υπέρ κατά αποχές δεκτές είναι οι ίδιες 60 και 61 υπέρ κατά αποχές δεκτές 62 και 22 ίδιες υπέρ κατά αποχές δεκτή 64 και 63. Διορθώνει ο πρόεδρος. Και άκρη 23. Υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτές. 63. Καταπίπτει αυτή. Πάμε στα εκτιμώντας. Πρώτη. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Τελική ψηφοφορία. Και όλο το κείμενο. Ηλεκτρονική ψηφοφορία παρακαλώ. Ψηφίζουμε τώρα. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας ψηφοφορίας. 57 υπέρ. 4 αποχές. Συγχαρητήρια. Ψηφίζουμε τώρα το νομοθετικό κείμενο με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Αρχίζει η ψηφοφορία. Ψηφίσαμε όλοι. Πέρας 5 57 ψήφοι υπέρ. Μία ψηφο. κατά. Τρεις αποχές. Συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια κύριε Σεγητά. Τελειώσαμε με αυτό. Περνάμε τώρα σε κάτι δυσκολότερο. Μια Ευρώπη που χρησιμοποιεί αποτελεσματικά τους σπόρους, σημείο 12, Χερμπραντή, ο συγητής. Πρέπει να συγκεντρωθούμε λίγο εδώ πέρα με τις ε, συμβιβαστικές ε, κάποιος ζητάει το λόγο. Πυρίλο, παρακαλώ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα είμαι σύντομος, αλλά νομίζω ότι πρέπει να σας επισημάνω κάτι που νομίζω ότι είναι σημαντικό. Δύο τροπολογίες υπέβαλα, την 22 και την 99, στα ισπανικά, εγγράφους. Ή στις μεταφράσεις της άλλες γλώσσες λέει το αντίθετο από αυτό που εγώ εσκόπευα να πω. Και δεν καταλαβαίνω πώς ακόμα και στα ισπανικά στα ισπανικά η, η μεταγραφή το πούμε λέει το αντίθετο επομένως παρακαλώ να διορθωθεί διότι λέει το αντίθετο από αυτό το οποίο ήθελα δεν ξέρω πώς αυτό θα διορθωθεί αλλά πρέπει να σας το πω και δεν καταλαβαίνω πώς είναι δυνατόν το, ε, το, το ισπανικό κείμενο τυπώθηκε στα ισπανικά και λέει το αντίθετο Ich würde vorschlagen, ich würde vorschlagen. Όταν θα έρθουν τα δύο αυτά σημεία σε ψηφοφορία, να διαβάσετε ξανά τις τροπολογίες σας και να το εξετάσουμε. Ε, συμφωνείτε, ωραία, έτσι θα κάνουμε. Για να μην χαθούμε στη μετάφραση. Ωραία, ξεκινάμε με την συμβιβαστική 1 ποιος είναι υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβιβαστική 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ενοποιημένη 6 υπέρ. Κατά. Αποχές να επαληθεύσουμε την συμβαστική 6. Ψήφισαν όλοι πέρας C6 απορρίπτεται περνάμε στην συμβαστική 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή συμβαστική 10 υπέρ κατά αποχές πρέπει να την εξετάσουμε παληθεύουμε λοιπόν την συμβαστική 10 άρχεται ψηφοφορία Σύρσαν όλοι πέρασε Συμβαστική 10 λοιπόν εγκρίνεται και συνεχίζουμε με την 11 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεν βλέπω από εδώ. Να επαληθεύσουμε λοιπόν τη συμβαστική 11. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Και αυτή γίνεται δεκτή. Συμβαστική 12 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 13 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Συμβαστική 15 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ κατά αποχές δεκτή περνάμε στην 1 τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 υπέρ κατά αποχές δεκτή 3 υπέρ κατά αποχές δεκτή 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή μετά θα πηδήξουμε μερικές ε, σελίδα 6 είμαι εγώ 57 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται προχωράμε πάλι παρακάτω Bei mir ist es die Seite 9. Σελίδα 9 και ψηφίζουμε την 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 91 υπέρ κατά αποχές δεκτή 93 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 95 υπέρ κατά αποχές δεκτή 92 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά Αποχές. Να επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά. Την 92. Μέρος πρώτο. άρχιε ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 36 υπέρ 23 κατά δεκτή. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 96 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ένα κατόπιν πάλι σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο ήτρε ένα υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά δεκτή. Αποχές δεκτή. 98. Πάλι σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 168. Καταπίπτη. 104 επίσης και ψηφίζουμε την 102 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 99 παρακαλώ άρα τον κύριο Περέλο να μας διαβάσει το κείμενο στη, στο πρωτότυπο Sí, gracias, señor presidente. Ε, ευχαριστώ. Λέει το κείμενο οποιαδήποτε δράση προς την κατεύθυνση το να γίνεται πιο αποτελεσματική χρήση των πόρων δεν είναι δυνατόν να περιοριστεί μόνο στον κρατικό δημόσιο τομέα διότι λέει, το λέει δηλαδή η μετάφραση ότι θα πρέπει να εξαιρέσει τον ιδιωτικό τομέα και να περιοριστεί μόνο στον κρατικό. Δηλαδή το αντίθετο αυτό που αποσκόπουσα να πω. Εντάξει, ε, δεν έχουν σημασία η λέξη και ακριβή διατύπωση, αλλά με το που λείπει κάποια λέξη έχουμε κείμενο που σημαίνει το αντίθετο. Να μην λέει επομένως μόνο στον κρατικό δημόσιο τομέα. Πράγματι σημαντική η διευκρίνηση. Ψηφίζουμε λοιπόν το κείμενο που μας διάβασε ο συνάδελφος. Αυτή είναι η 99 υπέρ. Κατά. Άποχες. Δεκτή ψηφίζουμε κατόπιν την 110 υπέρ συγγνώμη Wir müssen, Entschuldigung, abstimmen über... Συγγνώμη, ψηφίζουμε την 100. Οπότε ψηφίζουμε την υπαριθμόν 100 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 101 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 110 υπέρ κατά άποχες απορρίπτεται 111 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 112 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται να επαληθεύσουμε την 112 το μέρος δεύτερο ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας απορρίπτεται. Ίντα 10. Σε δύο μέρη πάλι. Μέρος πρώτο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 113 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή 114 υπέρ κατά αποχές δεκτή 115 υπέρ κατά αποχές δεκτή 119 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 121 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 116 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μέρος δεύτερο της 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτωται 120 υπέρ κατά αποχές δεκτή 143 υπέρ κατά αποχές δεκτή 122 υπέρ κατά αποχές δεκτή 123 υπέρ κατά αποχές δεκτή 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 127 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται όχι να ξαναδούμε την 127 127 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 128 υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 129 υπέρ. Σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται και να επαληθεύσουμε ξανά το δεύτερο μέρος άρχιδη ψηφοφορία. Haben alle abgestimmt. Πέρας. υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται το δεύτερο μέρος της 129. Παρακάτω. 38 σε τρία μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Μέρος δεύτερο της 38 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τρίτο μέρος υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την 88 υπέρ. Κατά. Αποχές, δεκτή. 133. Nein, wir müssen, wir müssen, zweiten Teil und den ersten Teil. Beide, ja? Okay, gut, wunderbar. Wir stimmen dann ab über, da müssen wir ein bisschen Text dringen, über Christas. Ψηφίζουμε την τροπολογία 240 της Κρίστα Κλάς. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Ήτρε 9. Όχι. Όχι, δεν χρειάζεται ψηφοφορία. 158 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 160 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 162 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 211 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 192 υπέρ κατά αποχές δεκτή 163 υπέρ κατά αποχές δεκτή 164 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 30 καταπίπτει 165 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 166 υπέρ κατά αποχές δεκτή 56 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 υπέρ κατά αποχές και έτσι έχουμε την τροπολογία που γίνεται δεκτή λοιπόν 177 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Ήτρα 6 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 10 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 202 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. Ήτρε 31 υπέρ κατά αποχές δεκτή ίντα καλύπτεται δεν ψηφίζεται 193 στην επόμενη σελίδα υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 194 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται μετά έχουμε τη 54 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 197 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται και θα την επαληθεύσουμε την 197 ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 32 υπέρ 25 κατά καλά κάναμε και το επαληθεύσαμε 203 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή τα 4 υπέρ κατά αποχές δεκτή ήτρε 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 207 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ συγγνώμη 205 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 204 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε την 204 άρχεται η ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. dafür, 32 26 υπέρ, 32 κατά. Απορρίπτεται. Να ε, δούμε τώρα την 206 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 210 υπέρ κατά αποχές δεκτή 212 υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε απορρίπτεται 213 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται το δεύτερο μέρος 214 υπέρ κατά αποχές 215 υπέρ κατά αποχές δεκτή το πρέπει οπότε περνάμε στην Ήτρε 20 υπέρ κατά αποχές δεκτή 21 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές Απορρίπτεται. 230 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 226 υπέρ. Ένας, μάλιστα. Κατά. Απορρίπτεται. 223 και 227 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 224 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.23 αποσύρεται δύο ταυτόσημες ε, μετά οι 2.29 και οι 2.22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.34 υπέρ κατά αποχές απορρίπτονται 2.28 υπέρ κατά αποχές δεκτή να, να την επαληθεύσουμε 2.28 ψήφισαν όλοι επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά την 2.28. Ψήφισαν όλοι. Πέρας. 31 υπέρ, 26 κατά, γίνεται λοιπόν δεκτή. Dann geht's weiter. 232 steht dann zur Abstimmung. Wer ist dafür? 2.32 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 2.31 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 2.35 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται, 2.36 Δεν ακούγονται τα γαλλικά. 2 ναι. 36 απορρίφθηκε και η 237 2.31 ε, και 2.35 με συγχωρείτε 2.36 ψηφίζεται τώρα Ποιο είναι υπέρ κατά αποχές να την επαληθεύσουμε ηλεκτρονικά 2.36 Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 25 υπέρ, 31 κατά. Απορρίπτεται. 237 υπέρ, κατά, αποχές, δεκτή. 16. Καταπίπτει. Και συνεχίζουμε με την 25 της Ήτρε. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 238. Σε δύο μέρη. Μέρος πρώτο υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. Μέρος δεύτερο υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 249 σε δύο μέρη. Δεν, δεν μου χρειάζεται. 2, 2.39 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Προχωράμε άρα παρακάτω στην τροπολογία του Ρίχα Τζέμπερ. 2.48 υπέρ κατά αποχές δεκτή. Είναι τα 8. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. Είναι τα 12. Υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 261 υπέρ. Κατά αποχές. Δεκτή. 262 υπέρ. Κατά αποχές. Απορριφθείτε. 263 υπέρ κατά αποχές να επαληθεύσουμε 263 με ηλεκτρονική ψηφοφορία η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρασε 31 υπέρ εγκρίνεται τα 5 υπέρ κατά αποχές δεκτή. τα 14 υπέρ, κατά αποχές δεκτή. τα 15 υπέρ, κατά όχι δεκτή. Συνεχίζουμε με την 265 χερπεράντι υπέρ κατά αποχές δεκτή 2 68 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 269 υπέρ κατά αποχές δεκτή 270 σε δύο μέρη μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.71 υπέρ κατά αποχές δεκτή 2.72 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 1 υπέρ κατά αποχές δεκτή είναι τα 9 υπέρ κατά αποχές δεκτή 6 υπέρ Judith Μέρκης, παρακαλώ. I have a, uh, uh, I have a Θέλω μία διευκρίνηση. Εκεί που λέει την τροπολογία 6, γιατί ακούσαν άλλε 3, ήταν κάποια ομαδική ψηφοφορία. Δεν θέλω να ρωτήσω τη γραμματεία γιατί η 88 θεωρείται ότι καλύπτει την, και την 133. Δεν συμφωνώ. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει χωριστή ψηφορία για την 133. Ίσως δηλαδή το τελευταίο τμήμα καλύπτεται, αλλά το πρώτο τμήμα όχι. Άρα γίνεται να ψηφίσουμε το πρώτο τμήμα της 133. Πρόεδρος. Εγκρίθηκε 88, οπότε δεν ε, έχει πια νόημα. Έτσι μου λένε εδώ πέρα ότι τα κάναμε κανονικά τα πράγματα. Εντάξει, συνεχίζουμε με την παριθμόν 6 υπέρ κατά αποχές δεκτή 7 υπέρ κατά αποχές δεκτή 8 υπέρ κατά αποχές δεκτή 9 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 10 υπέρ κατά αποχές θα την επαληθεύσουμε την υπαριθμόν 10 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 31 υπέρ 25 κατά 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 μέρος πρώτο υπέρ κατά αποχές δεκτή μέρος δεύτερο υπέρ κατά αποχές δεκτή 12 μέρος α καταπίπτει δεν χρειάζεται να την ψηφίσουμε γιατί αυτή είναι 14 15. είναι προσθήκη και πρέπει να την ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε την 15 υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 16 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 17 υπέρ κατά αποχές δεκτή 18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα επαληθεύσουμε για να είμαστε σίγουροι την 18 άρχεται η ψηφοφορία ψήφισαν όλοι πέρας 25 υπέρ, 29 κατά. Απορρίπτεται. 19 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 20 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 21 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 22 υπέρ. Α, 22 ο κύριος Πυρίλα διευκρινίστε παρακαλώ για να ξέρουμε τι θέλετε ακριβώς. Διαβάστε λοιπόν το πρωτότυπο. Pues con toda rapidez, señor presidente. Σύντομα ε, ε, σας διαβάζω ε, το κείμενο που λέει, που έχει προσθεθεί και λέει, από εκεί που λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση ότι εν πάση περιπτώσει δεν είναι δυνατόν να προχωρήσουμε προ την βιωσιμότητα, την εφορία, χωρί να υπάρχει εμπλοκή εκείνων, δεν εννοεί του πολίτε, μέσω μια αλλαγή νοοτροπία και επίση μια αλλαγή των συνδυών τη κοινωνία σε σχέση με την χρήση των πόρων. Gut, jetzt haben wir den την Μάλιστα τώρα έχουμε το πρωτότυπο κείμενο, είναι σαφέ και το ακούσατε. Ψηφίζουμε λοιπόν τροπολογία 22. Ποιοι είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Δεκτή. 23 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται 24 υπέρ κατά αποχές δεκτή 25 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 26 υπέρ κατά αποχές δεκτή 27 Α, ζητάτε επανέλεγχο τις 26 μάλιστα άρχεται η ψηφοφορία Ψήφισαν όλοι. Πέρας. Απορρίπτεται. Η 26. 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Υπάρχει ένα λάθος εδώ πέρα στον κατάλογο. Υπάρχει προφανώς ένα μόνο συμπέρασμα και μία μόνο τελική ε, ψηφοφορία. Οπότε θα ψηφίσουμε τώρα μία και καλή για την ε, έκθεση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Λείπουν ακόμη τρεις. Δεν θέλουν να ψηφίσουν. Ωραία, πέρας. 48 υπέρ τρεις ψήφοι κατά, πέντε αποχές συγχαρητήρια στον κύριο Γερμπραντή για την έκθεση αυτή πρωτοβουλίας. Ε, ευχαριστούμε, ευχαριστούμε και τη γραμματεία. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Δοκιμάζονται τα νεύρα. Και συνεχίζουμε στην έκθεση Ζανόνι, γνωμοδότηση. Das ist der ehemalige 13, der Το θέμα το οποίο αφορά τροποποίηση του κανονισμού ΤΑΔΕ σχετικά με την αφαίρεση πτερυγίων καχαρία επί του σκάφους. Ξεκινάμε με την τροπολογία 6 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 7 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 8 υπέρ. Κατά. Ε, υπέρ, με Κατά. Αποχές δεκτή. 9 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. 10 υπέρ. Κατά. Αποχές δεκτή. Αιτιολογικές σκέψεις. 11 υπέρ κατά αποχές δεκτή εκτιμώντας 12 υπέρ κατά αποχές δεκτό 13 υπέρ κατά αποχές δεκτή 14 υπέρ κατά αποχές δεκτή 15 υπέρ κατά αποχές δεκτή 16 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 17, 3 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 17 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 4 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 18 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή. 5 υπέρ. Κατά αποχές δεκτή και ψηφίζουμε τώρα ολόκληρη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής μας για το θέμα αυτό με ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Πέρασε. 50 υπέρ, 2 κατά, καμία αποχή και εγκρίθηκε άρα η γνωμοδότηση αυτή. Σας ευχαριστώ για τη συγκέντρωσή σας. Τελειώσαμε με τις ε, ψηφοφορίες και όσοι θέλουν να μείνουν, καλώς να μείνουν. Ε, στους υπόλοιπους καλή σας ημέρα. Περνάμε τώρα στο σημείο υπαριθμών 15 της ημερήσιας διάταξης εκτελεστική πράξη για τις ζωοτροφές και τα τρόφιμα από την Ιαπωνία μετά το ατύχημα στη Φουκουσίμα. Wir begrüßen heute ε, σας παρακαλώ, μπορούμε λίγο να, να συζητήσουμε. Ε, ή δεν θέλετε περάστε έξω. Έχουμε λίγη ώρα μέχρι να έρθει ο Επίτροπος, οπότε θα ήθελα να περάσουμε σε αυτό το θέμα. Καλωσορίζω μια Ιαπωνική αντιπροσωπεία εδώ στην αίθουσα. Καλώς ήρθατε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θα δώσω τον λόγο στον κύριο Πουντελέ από την Κομισιόν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα. Σύντομα δύο λόγια για το ιστορικό πλαίσιο. Θα θυμάστε όλα συνέβη το ατύχημα στη Φουκουσίμα αντέδρασε ταχύω η Κομισιόν, ώστε να λεφθούν κάποια μέτρα για να υπάρξει κάποιο έλεγχο τη ε, ραδιενέργεια επί των τροφίμων στην Ιαπωνία. Λάβουμε αυτά τα κατεπήγοντα μέτρα τότε, ούτω ώστε να μπορέσουμε ε, να έχουμε το νομικό πλαίσιο και το τεχνικό και τα κράτη-μέλη να μπορέσουν να ελέγξουν την εισαγωγή για ό,τι προϊόν εισήγεται από την Ιαπωνία και βασικά έχουμε διάφορα φυτικά προϊόντα που εισάγουμε ε, φύκια, λαχανικά, τέτοιου είδου φυτικά προϊόντα επίσης ε, προϊόντα αλλιεία όχι κρέας όμως ούτε γαλακτοκομικά επίσης εισάγουμε μικρές ποσότητες ζωοτροφές για, για οικιακά ζώα και έτσι επομένως ε, θεσπίστηκαν ε, αυτοί, αυτοί οι ευρωπαϊκοί κανόνες της εποχής του Τσερνομπίλ για να μπορεί να ασκείται έλεγχος και επίσης οι Ιάπωνες Έχουν και αυτοί και δικούς τους βέβαια κανόνες όσον αφορά τον έλεγχο αυτών των εξαγωμένων προϊόντων. Και έτσι έχει επιβληθεί αυτή η υποχρέωση για τις αρχές της χώρας τους, ώστε να κάνουν τέτοια, τέτοιους ελέγχους πριν εξαχθούν τα προϊόντα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καλύπτονται συγκεκριμένε περιοχές και είπαμε ότι είναι 100% έλεγχος εκεί και είναι ψηλό ποσοστό του ελέγχου ή στην άφηξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη. Έγινε συζήτηση στο Κοινοβούλιο, όπως θα θυμάστε, και επίσης και στην Ολομέλεια στο Στρασβούργο στις 8 Τετάρτου του 11. Και τότε το Κοινοβούλιο απίτησε να αλλάξει το νομικό καθεστώς ούτως ώστε να προσαρμοστεί στις αυστηρότερες ιαπωνικές διατάξεις Επομένως, κατόπιν αυτή τη συζήτηση και εμεί τροποποιήσαμε τις σχετικέ διατάξεις, ώστε να επικαλούμεθα τις ιαπωνικές αυστηρότερες ε, διατάξει. Και από την 1η Απριλίου οι Ιάπωνε αναβάθμισαν το νομικό καθεστώ και είναι ακόμη αυστηρότερο τώρα ούτω ώστε να ανακτήσουν την εμπιστοσύνη των καταναλωτών. Είχαμε επομένω την επιλογή ή να κρατήσουμε τις παλαιότερες διατάξεις ή να προσαρμοστούμε στις νέες, αυστηρότερες ιαπωνικές. Και επειδή θέλαμε να είμαστε συνεπείς, για να αποφύγουμε το να έχουμε τις πιο αυστηρές ιαπωνικές διατάξεις ε, ε, για τους ελέγχους των προϊόντων τους πριν την εξαγωγή και εμείς όταν κάνουμε τον έλεγχο εδώ ε, άμα αφήξει να έχουμε επικέστε διατάξεις για να είμαστε συνεπείς προτείναμε να αναβαθμιστούν οι διατάξει, να γίνουν αυστηρότερε και να ταυτιστούν με τις ε, Ιαπωνικές και γι' αυτό το λόγο τον Μάρτιο προτείναμε στα κράτη-μέλη ένα σχέδιο κανονισμού μα, ούτω ώστε να προσαρμοστούμε στι νέες αυστηρότερες Ιαπωνικές διατάξεις. Επίσης, με την ευκαιρία αυτής της αποφάσεως θελήσαμε να προσαρμόσουμε τους ελέγχους για το ιαπωνέζικο ουίσκι, το σακέτα, τα, τα αλκοολούχα, τα ιαπωνικά, διότι οι Ιάπωνες προχώρησαν σε θέσπιση κάποιων αναλύσεων για αυτά τα ποτά, τα οποία σε μικρές ποσότητες εξάγουν προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν υπήρχε πρόβλημα διότι η διαδικασία της ορίμανσης, της, της απόστασης κλπ. Εάν υπήρχε περίπτωση μόλυνσης από την ραδιενέργεια, ας πούμε από τα σιτηρά που χρησιμοποιούνται για να παραχθούν αυτά τα ποτά, αν υπήρχε επομένω τέτοια μόλυνση, τότε θα έμενε στα κατάλοιπα τα οποία δεν μπαίνουν στο, στο, στο ενόπνευμα γιατί μέσω της απόσταξης η ραδιενέργεια δεν περνάει στους, ε, στους ατομούς που κατόπιν μετά με κάποιο είδους ε, στερεοποίηση, υγροποίηση γίνεται σούτσου, σακέ, αυτά τα ποτά τέλος πάντων. Οπότε, επί τη βάση αυτών των ε, στοιχείων και των ελέγχων των Ιαπώνων προτείναμε στα κράτη-μέλη αυτά τα τρία ποτά να εξαιρεθούν από τους ελέγχους στο σημείο εισαγωγή στην Ευρωπαϊκή Ένωση οπότε. Ε, κάτι επιγόντως ελήφθη για αυτή η τρίτη απόφαση γιατί θέλουμε να είμαστε συνεπείς σε σχέση με την Ιαπωνική απόφαση της αλλαγής του νομικού πλαισίου την 1η Απριλίου και για αυτό και εμείς κατεπηγόντως λάβουμε αυτή την απόφαση πριν απαντήσω στις ερωτήσεις που τυχόν έχετε, θα πρέπει να σας πω ορισμένα αριθμητικά στοιχεία. Οι Ιαπωνικές αρχές έχουν κάνει από τότε που συνέβη το στην ε, Φουκουσίμα 136.000 αναλύσεις όσον αφορά τα τρόφιμα εκεί, στην Ιαπωνία, όσον αφορά την εσωτερική κατανάλωση και από την 1η Απριλίου με το νέο νομικό πλαίσιο το αυστηρότερο έχουν κάνει 8.000 συνολικά 1.380 ελέγχους όσον αφορά το ουίσκι, το σακέ και το σότσου χωρίς να επισημανθούν ίχνη ραδιενεργίας. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση τώρα, Άμα τη εισαγωγή για αυτά τα προϊόντα, για αυτά τα τρόφιμα, οι αρχές μας έκαναν από πέρσι, από τον Μάρτιο, από τον Μάρτιο του 2011, σχεδόν 2.000 ελέγχους μέσα στο 2011 και 500 ελέγχους το 12 φέτος. 2.500 και διαπίστωσαν δύο φορές ότι υπήρχε πρόβλημα ε, δύο φορές σε περιπτώσεις ε, τσαγιού σε φύλλα. Αυτά, αν θέλετε διευκρινήσεις ή αν έχετε υποβάλλετε ερωτήσεις, ευχαρίστως να σας απαντήσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τις πληροφορίες σας, Κομισιόν. Μια πρώτη παρατήρηση. Ξέρετε ότι εμείς οι Ευρωβουλευτές δεν συμφωνούμε αρκετά με αυτή τη διαδικασία. Ο κύριος Λάινεν έστειλε μια επιστολή που έλεγε ότι θα πρέπει η Κομισιόν να μας δώσει από την αρχή της πληροφορία. Ενώ εσείς ενεργήσατε χωρίς να γνωρίζουμε εμείς τίποτα. Ζητώ συγγνώμη, αλλά δεν νομίζω ότι είναι σωστά όλα αυτά. Το παίζετε μοναχικός καβαλάρης, όπως λέμε εμείς στη Γαλλία. Δεν είναι σωστό αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά το περιεχόμενο της πρότασης. Ακόμα και σήμερα πρέπει να πούμε το εξής, κύριε Πουντλέ. Έχουμε αρκετές αβεβαιότητες για τους τέσσερις αντιδραστήρες. Ε, οι τρεις έχουν α, λιώσει και στον τέταρτο έγινε μία έκρηξη και έχουμε και αμερίκιο και πλουτόνιο και κέσιο που εκλείεται γύρω από τον αντιδραστήρα. Ένας Αμερικανός γερουσιαστής έστειλε μια επιστολή που μας λέει ότι είναι πολύ ανήσυχος για την κατάσταση του αντιδραστήρα. Και θέλω μάλιστα επευκαιρία να ζητήσω από την Κομισιόν να γίνει μια ευρωπαϊκή αποστολή με ευρωβουλευτές, αλλά και με μέλη της Κομισιόν και ενδεχομένως, γιατί όχι, μέλη από τα κράτη-μέλη. Για να κάνουμε, λοιπόν, μια αποστολή επιτόπου στη Φουκουσίμα. Εγώ πήγα, αλλά ήμουνα πέρα από τα 60 χιλιόμετρα, έτσι, που ήταν ούτως ή άλλως πολύ μολυσμένη, αλλά δεν έφτασα στο επίπεδο βέβαια του αντιδραστήρα. Όταν βλέπουμε τι παραπληροφόρηση η ΤΕΠΚΟ και οι Ιαπωνέζικες αρχές, νομίζω ότι είναι ανησυχητικά όλα αυτά και καλό θα ήταν να πάμε να δούμε τι γίνεται, γιατί πιστεύουμε ότι ακόμα υπάρχει έκκληση ραδιενέργειας. Και τώρα πάω στο τρίτο στοιχείο. Λέτε τώρα ότι τώρα δεν έχουμε να ε, λόγο να μετρήσουμε το στρόντιο, το ιόδιο και το αμερίκιο. Αυτά τα τρία δεν χρειάζεται να τα μετράμε. Είναι πολύ νωρί νομίζω να σταματήσετε αυτού του τρει ελέγχου. Γιατί Σποραδικά υπάρχουν εκκλήσεις, ε, υπάρχει ραδιενέργεια γύρω από το χώρο των πυρηνικών εγκαταστάσεων. Ε, ούτως ή άλλως δεν έχουμε την άδεια να πάμε στο χώρο της πυρηνικής ε, εγκατάστασης. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους κανόνες. Νομίζω ότι είναι απίστευτο, γιατί είχαμε ψηφίσει και ξέρετε ότι οι οικολόγοι είχαν πει ότι οι κανόνε σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματος που καθορίζονται από την Κομισιόν και επομένω από του εμπειρογνώμονες τη Euratom ήταν πολύ αυστηροί. Είχαμε φτάσει στα 1000 μπεκερέλ το κιλό για το κέσιο. Ούτως ή άλλως σε λίγες μέρες θα ξεπεράσουμε την μέγιστη αποδεκτή δόση. Και μου είπαν όχι, όχι, όχι. Γίνεται το ατύχημα της Φουκουσίμα και το επίπεδο των Ιαπωνέζων ήταν στο μισό, 500 μπεκερέλ. Ζητήσαμε λοιπόν μία ευθυγράμμιση από τον κύριο Μπαρόζο. Πρέπει να ευθυγραμμιστούμε ε, με τους Ιαπωνέζους, γιατί δική μας κάνουν ήταν η διπλάση από τους Ιαπωνέζους. Και τώρα φτάσαμε ακόμα πιο κάτω, 100 μπεκερέλ και 10 μπεκερέλ. Επομένως, τώρα το, εξι... Ε, το εξή πρόβλημα. Γιατί εισάγουμε Ιαπωνέζικα προϊόντα, αν μου πείτε, στο ουίσκι, στο σακέ. Δεν υπάρχει ραδιενέργεια. Οκ, εντάξει, με την απόσταξη δεν περνάει το κέσιο. Αλλά για τον τρίτιο δεν ισχύει αυτό. Εγώ έχω ένα εργαστήρι ε, μέτρησης της ε, ραδιενέργειας. Υπάρχουν κάποια ραδιονουκλείδια που δεν περνάνε, κάποια άλλα που περνάνε. Οι μετρήσεις που έγιναν για αυτά τα αλκοολούχα ποτά έγιναν τους Ιαπωνέζους. Θα πρέπει να μετρήσουμε όλα τα ραδιονουκλεΐδια. Σε ό,τι αφορά το τσάι. Ξέρετε, ότι δύο δείγματα τσαγιού ξεπέρασαν τα 500 μπεκερέλ το κιλό. Και λέτε, ναι, αλλά είναι, υπάρχει μια διάλυση και τα ποσά που βρήκαμε δεν είναι σοβαρά. Κι όμως είναι, είναι πολύ σοβαρό το θέμα, γιατί η θεωρία είναι ότι οποιαδήποτε δόση ραδιενέργειας μπορεί να ε, δημιουργήσει, να αυξήσει τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου. Γιατί κάποιος ο οποίος πίνει το γιαπωνέζικο τσάι του με 10 μπεκερέλ, α πούμε, και Ε, γιατί να το πιει, δηλαδή, αν θα μπορούσε να πιει ένα τσάι με 0 μπεκερέλ κεσίου. σίου. Ποιο είναι το, ο λόγο που εισάγουμε γιαπωνέζικο τσάι, ενώ μπορούμε να εισάγουμε τσάι με 0 μπεκερέλ. Γιατί να εισάγουμε γιαπωνέζικα προϊόντα, λοιπόν, για οικονομικού λόγου. Υπάρχει ένα θέμα όμως υγείας εδώ. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε αυτό που κάνει η Αυστραλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε. Σταμάτησαν τι εισαγωγέ Ιαπωνέζικων προϊόντων. Δεν νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό οικονομικά για τους Ιαπωνέζους, αλλά από την άλλη είναι πολύ σημαντικό για την ε, υγεία των Ευρωπαίων και γινόμαστε πολύ πιο αξιόπιστοι. Επαναλαμβάνω, θέλω επίσημα να ζητήσω από την Κομισιόν να γίνει ε, αποστολή στην ε, Ιαπωνία, στη Φουκουσίμα, για να δούμε τι γίνεται. Ποια είναι η κατάσταση των δραστήρων, τι εκλείεται από τους αντιδραστήρες αυτούς. Δεύτερον, ζητά από την Κομισιόν να μας επανεξιολογήσει τους κανόνες, γιατί βλέπω ότι οι κανόνες μας ήταν πολύ πιο ψηλά και άρα πιο χαλαροί. Ε, καλό είναι να κατεβάζουμε τα όρια σε περίπτωση πυρηνικού ατυχήματο και τρίτον, να σταματήσουμε τις αγωγές πονέζικων προϊόντων. Γιατί δηλαδή να εισάγουμε ραδιενέργεια στην Ευρώπη. Γιατί να είμαστε τόσο δημοκρατικοί στη ραδιενέργεια. Υπάρχει κανένα λόγο. Ευχαριστώ. Ιβ Κοσέ. Ο επόμενος ομιλητής. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα είμαι πιο σύντομος, γιατί η κυρία Ριβαζή με κάλυψε σε μεγάλο βαθμό. Να συμπληρώσω την παρέμβασή της και τα ερωτήματα προς την Κομισιόν. Από τη μία, ήρθε ο παλιός νομάρχης της ε, περιοχής της Φουκουσίμα, που ήταν νομάρχης για 16 περίπου χρόνια, ήρθε στην Ευρώπη λοιπόν και μας είπε με ποιους δύσκολους όρους ε, ζουν εκεί οι γεωργοί. Ε, πριν από τρεις εβδομάδες, ε, ένα μήνα, ήρθα σε επαφή με έναν γεωργό που μου είπε ότι λόγω τη ραδιενέργεια δεν μπορεί πια να πουλήσει την γεωργική παραγωγή του. Είχαμε και εμείς αυτή την πληροφόρηση, την ανησυχητική, ότι το πράγμα συνεχίζεται, δεν έχει σταματήσει. Φυσικά, μπορούμε να κατεβάσουμε τους κανόνες για τα τρόφιμα, αλλά τα πράγματα είναι διαφορετικά το Τσερνομπίλ. Εκεί έγινε μια τεράστια έκρηξη και μετά μέσω του συνέφου ας πούμε έστειλε παντού στην Ευρώπη τα ραδιονουκλεΐδια. Ας τα πούμε ειλικρινά τα πράγματα, αλλά στη Φουκουσίμα το πράγμα κρατάει πολύ καιρό. Είναι ένας πυρηνικός πόλεμος χωρίς να υπάρχει χωρίς να γίνεται πόλεμο στην πραγματικότητα. Δηλαδή, τι θέλω να πω, ότι συνεχίζεται το πρόβλημα στην πισίνα, το πουλ αυτό του τετάρτου αντιδραστήρα. Γι' αυτό αυτό που λέει η κυρία Ριβαζή να το ακούσει η Κομισιόν και το Κοινοβούλιο, για να πάμε να δούμε τι γίνεται με αυτή την πισίνα του τέταρτου αντιδραστήρα, του αντιδραστήρα υπαριθμών 4. Όπως η κυρία ε, Ριβαζή, ε, θέλω να πω ότι υπάρχει το ΣΕΡΕΜΕΣ, ένα ανεξάρτητο εργαστήριο α, στη Γαλλία για τη ραδιενέργεια, 25 χρόνια μετά το Τσερνομπίλ, πρέπει να έρθουμε σε επαφή με αυτό το εργαστήρι. Πρέπει να έρθουμε σε επαφή με την κοινωνία των πολιτών. Ε, εντάξει, έχουμε τους εμπειρογνώμονες. Αλλά θα πρέπει και το CRMS, αυτό το εργαστήριο, ε, και άλλοι φορείς της κοινωνίας των πολιτών, αν γίνει αυτή η αποστολή, να έρθουν αυτοί σε επαφή με τους επίσημους ε, εμπειρογνώμονες. Δηλαδή, το CRMS να έρθει σε επαφή με επίσημου εμπειρογνώμονες. Ευχαριστώ. Κύριο Σπακ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεν θα είμαι πολύ φλίαρος, δεν θα μακρηγορήσω. Θα ήθελα να πω στην Κομισιόν ότι το ΣΑΚΕ παράγεται με ζήμωση και όχι απόσταξη. Ζήμωση. Και επομένως, αν θεωρείτε ότι η απόσταση ε, σημαίνει ότι το, ότι το ΣΑΚΕ είναι ασφαλές, κάνετε λάθος. Επίσης, Κομισιόν, έχετε τίποτα μοντέλα για την εξάπλωση της ε, ραδιενέργειας της θάλασσας γύρω από την Ιαπωνία. Ευχαριστώ, Παύλ Πακ. Και τώρα θα μας μιλήσει ο κύριος Πουλέ, να λάβει το λόγο για να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Δεν έχω αρμοδιότητα τόσο ώστε να σας φτιάξω μια τέτοια αποστολή προ την Ιαπωνία, αλλά τέλο πάντων θα, θα, θα διαβιβάσω το έτοιμά σα, κυρία μου, Αρμοδίω, κανένα καμία εντύπωση. Δεν ξέρω πώ αυτό θα μπορούσε να οργανωθεί. Θα μιλήσω πάντω με τη Γενική Γραμματεία, του συναδέλφου τη Γενική Διεθνή για την Ενέργεια, εκείνοι που ασχολούνται με τα πρότυπα αλλά και με το περιβάλλον. Κανένα πρόβλημα. Τώρα, όσον αφορά τα άλλα ραδιοστοιχεία, γνωρίζετε ότι το ιόδιο έχει ημιζωή οκτώ ημερών. Δηλαδή 8 μέρες μετά το πρόβλημα της μόλυνσης, το ιόδιο κατά το ίμιση ξαφνίζεται και μετά στη συνέχεια. Όποτε στην αρχή έγινε αυτός ο έλεγχος, ζήτησα από τα κράτη-μέλη να κάνουν έλεγχο και κατόπιν προέκυψε ότι δεν χρειαζόταν ανάγκη ελέγχου και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να σταματήσουν το στην επικεντρώσει προσπαθειές τους Justo Chiesio. De 3 ans et le 137 qui a une durée 30 ans, Το 134. Γιατί έχει μια ζωή 80 ετών. Οπότε από τη αυτών προέκυψαν κάποια στοιχεία. Σύμφωνα τα οποία υπάρχει μόλυνση, αλλά είναι ελαφρότατη. Πολύ μικρή. Και επειδή οι αρχές των 11 πληγισών περιοχών προβαίνουν σε 100% έλεγχο των εξαγωγών, κάνουν εκείνη τον έλεγχο και είπαμε ότι εμείς δεν χρειάζεται να το κάνουμε. Διότι είπαμε ότι εμπιστευόμαστε τις Ιαπωνικές αρχές, ίσως αυτό το θεωρείται συζητήσιμο, αλλά εμείς τους εμπιστευτήκαμε. Και επί τη βάση αυτής της εμπιστοσύνης, ε, άλλωστε έχουμε μια έκθεση με όλο το αποτέλεσμα των ελέγχων των 138.000 και τόσο, τόσο ελέγχων. Ούτω ώστε μπορούμε να παληθεύσουμε. Τώρα, για το τσάι. Εισάγουμε τσάι από την Ιαπωνία. Βεβαίω και θα πρέπει να ασκείται έλεγχο στις αγωγέ. Αλλά έχουμε πολύ αυστηρότερες διατάξει. Ε, από ότι για το Τσερνομπίλ. 1150 και άλλοι έχουν 500. Δηλαδή εμείς, εμείς έχουμε διπλάσιο, διπλάσιο και όριο σε Μπεκερέλ. 1250 από 500. Και πρόκειται για το πράσινο τσάι σε φύλλα χήμα. Και ε, μπαίνει βέβαια ζεστό νερό. Εν πάση περιπτώσει είναι όμως πολύ αυστηρότερε οι δικές μας διατάξει. και κάνουμε την εισαγωγή γιατί έχει καλή φήμη το, το, το, το τσάι αυτό. Για, κοιτάξτε, δεν υπήρχε πολιτική βούληση να απαγορεύσουμε όλες τις εισαγωγές. Λήφθη η πολιτική απόφαση να κάνουν πιο αυστηρέ τι διατάξει και του ελέγχου και να ζητήσουμε από του Ιαπωνέζου να κάνουν 100% έλεγχο με την εξαγωγή. Και τα κράτη-μέλη 5, 10 και 20% ανάλογα με την περίπτωση, ανάλογα με το προϊόν, να ασκούν έλεγχο ε, άμα τη εισαγωγή, ούτως ώστε να επαληθεύεται κατά πόσον η έλεγχη η, η είναι αξιόπιστη. Να επαληθεύσουμε δηλαδή, να επαληθεύσουμε ότι όντω είναι αξιόπιστη η Ιαπωνική έλεγχη. Οπότε όλα τα στοιχεία που σήμερα έχουμε καταδεικνύουν το ότι ναι, μπορούμε να εμπιστευόμαστε τους Ιάπωνες όσον αφορά αυτούς τους έλεγχους. Τώρα, όσον αφορά τους αντιδραστήρες. Εμείς είμαστε ειδικοί στα είδη διατροφής, στα τρόφιμα, όχι στην ε, ραδιενέργεια, αλλά οι συνάδελφοι της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργεια και Περιβάλλον ε, βοηθούμενοι και από την ε, Διεθνή Αρχή Ατομικής Ενεργείας πήγαν επί τόπου, ε, επιθεωρητές, ελέγξανε και είπαν ότι σταθεροποιήθηκε η κατάσταση τους αντιδραστήρες. Υπήρξαν διαρροές, ναι. Κανείς δεν το, δεν το, το αρνείται αυτό, ούτε οι, οι αρχές της χώρας. Σήμερα όμως θεωρείται η κατάσταση σταθερή. Εάν τώρα επιδεινωθεί η κατάσταση, εάν έχουμε καινούργιες εκρήξεις, ε, τότε θα ξαναλάβουμε τα μέτρα μας και όπως το παρελθόν θα κάνουμε ότι, ό,τι κάνουμε δηλαδή μέσα σε 48 ώρες. Θα ενισχύσουμε τους νόμους, θα απαγορεύσουμε, θα, θα, θα, θα αλλάξουμε τις κανόνες για τα για τα ίχνο στοιχεία αυτά, το πλουτόνιο δηλαδή, εάν μαζικά μολύνει το περιβάλλον, ε, μπορούμε μέσα σε 24-48 ώρες να αλλάξουμε τις διατάξεις και να προσθέσουμε στα, στις περιορισμούς το πλουτόνιο. Κανένα πρόβλημα Τώρα, έχουμε λάβει τη διαβεβαίωση ότι έχει σταθεροποιηθεί η κατάσταση στους αντιδραστήρες, σε εκείνους που πριν από ένα χρόνο είχαν εκραγεί. Τώρα, επαναξιολόγηση των διαταξιών μας, αυτό ξέρετε ότι είναι θέμα της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας. Είναι η ειδική του άρθρου 31, έτσι τους λέμε, Αυτή που είναι ειδικοί σαν ατομική ενέργεια και είναι εκείνοι που ασχολούνται με την αναθεώρηση των σχετικών διατάξεων, για να προσαρμόσουν, να τροποποιήσουν τις σχετικές διατάξεις αυτές που θεσπίστηκαν τότε με το Τσερνομπίλ προ 20 ετίας που παρέχουν θεωρητικά λιγότερη προστασία. Τώρα και να απαντήσω στον κύριο Κωσέ όσον αφορά τη χρησιμοποίηση ανεξαρτήτων εργαστηρίων χρησιμοποιούμε όλα τα στοιχεία που μας διάθεσή Πήγε η Greenpeace, πήρε δείγματα, έκανε αναλύσεις επιτόπου ή αλλού και εμείς λαμβάνουμε υπόψη όλες αυτές τις αναλύσεις όσον αφορά την τεχνική ανάλυση του τι ισχύει επί τόπου. Και αν γίνει μια τέτοια κοινή αποστολή μεταξύ ημών και ημών, εντάξει, δεν μπορούμε εμείς, εμείς όμως να, την οργανώσουμε ή να φτιάξουμε το πρόγραμμα της αποστολής. Είναι όμως πάρα πολύ καλή ιδέα. Να πάμε να δούμε τι γίνεται. Κύριε για το ΣΑΚΕ, ναι. Η παλαίωση και η απόσταξη και η ζήμωση. Φιλτράρεται στη, για, τη ζήμωση για του ΣΑΚΕ, φιλτράρονται τα στερεά στοιχεία και χρησιμοποιούνται τα υγρά. Και από ό,τι μας λένε, σύμφωνα τα τεχνικά στοιχεία, λένε οι Ιαπωνέζοι ότι αν υπάρχει ραδιενέργεια στο ρύζι, αυτή η ραδιενέργεια μένει στα στερεά, δεν περνάει ή στα υγρά. Επίσης, βγάζουν το φλοιό του ρυζιού, το υπόλοιπο είναι γυαλισμένο και εν πάση τόση, αυτός ο φλοιός, το εξωτερικό, το εξωτερικό κομμάτι του ρυζιού έχει τη ραδιενέργεια. Α, αυτά πρόεδρε για να απαντήσω όσα ζήτησαν οι βουλευτές. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εμείς ευχαριστούμε, κυρία, για τις απαντήσεις σας, για τις απαντήσεις, για τις... Και τώρα ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με τον ε, Επίτροπο για τα θέματα υγείας. Θα κάνουμε ανταλλαγή απόψεων. Βλέπω πάρα πολύ σηκώνει το χέρι. Πάρα πολύ συνάδελφοι, ακριβώ αυτό δείχνει τον ενδιαφέρον για την ανταλλαγή απόψεων και αυτό διότι φέτο αλλά και του χρόνου έχουμε μία σειρά νομοθετημάτων που ετοιμάζονται. Και θα ακολουθήσουμε την πάγια διαδικασία, δηλαδή θα έρθει ο Επίτροπος να μας παρουσιάσει το τι γίνεται, δηλαδή 10 λεπτά και 100 θα έχουμε δύο ή 3 γύρους ερώτα απαντήσεων. Επομένως, να μην αναλώνουμε περαιτέρω το χρόνο που έχουμε και έχετε σκητάλη αυτής αμέσως κύριε Πρόεδρε για τη δήλωσή σας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, είμαι πολύ χαρούμενος που εμφανίζομαι στην Επιτροπή σας για τον τρίτο διαρθωμένο διάλογο ως Επίτροπος Υγείας και Πολιτικής Καταναλωτών. Θα ήθελα να ξεκινήσω ευχαριστώντας τον κύριο Τζολί για την καλή συνεργασία που είχαμε ε, όσο καιρό ήταν πρόεδρος αυτής της Επιτροπής εδώ περιβάλλοντος. Και ελπίζω να έχουμε το ίδιο επίπεδο συνεργασίας και διαλόγου σε αυτό το δεύτερο μισό της κοινοβουλευτικής θητείας με τον νέο πρόεδρο. Θα ήθελα να σας πω από την αρχή ότι μου είναι πολύτιμη η συμβουλή και η συνεισφορά σας, εσάς των μελών τη επιτροπή του περιβάλλοντο. Όλε οι συμβουλέ που μου δώσατε στο παρελθόν τις έλαβα υπόψη μου και ελπίζω να συνεχίσουμε την ίδια επιτυχή συνεργασία. Θα ήθελα να σταθώ σε μια σειρά από θέματα που ενδιαφέρουν ιδιαίτερα στην Επιτροπή σα αυτή την παρουσία μου εδώ και κυρίω αυτά τα οποία είναι τώρα υποσυζήτηση ή που έχουν δρομολογηθεί για να συζητηθούν στο εγγύς μέλλον. Φυσικά δεν υπάρχει περίπτωση να καλύψω όλα όσα σας ενδιαφέρουν σε αυτή την σύντομη πανεβασή μου. Καταρχάς γιατί έχετε ένα τεράστιο εύρος θεμάτων που σας απασχολούν. Έχετε μια μεγάλη εντολή. Αλλά πιστεύω ότι θα έχουμε πολλές ευκαιρίες να θέσουμε και άλλα θέματα στο, στη φάση ρωταποκρίσεων που ακολουθεί. Να ξεκινήσω με κάποια θέματα που είναι εξελίξη. Το πρόγραμμα υγείας για την ανάπτυξη. Καταρχάς, το νέο αυτό πρόγραμμα Υγεία για την Ανάπτυξη θα εξυπηρετήσει ή θα μας δώσει πραγματική ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία και θα ενισχύσει περισσότερο τη σχέση ανάμεσα σε έναν υγιή πληθυσμό και στην οικονομική ανάπτυξη. Να πω κάτι σημαντικό εδώ. Η Κομισιόν πρότεινε το μελλοντικό πρόβλημα που θα ονομάζεται Υγεία για την Ανάπτυξη. Το πρότεινε γιατί η υγεία είναι ένας είναι μια πολιτική από μόνη της. Και ο στόχος μας είναι η επίτευξη της υγείας. Ορισμένοι από εσά θεωρούσαν ότι ο τίτλος σημαίνει ότι η υγεία ε, είναι δευτερογενή σε σχέση με την ανάπτυξη. Όχι, σε καμία περίπτωση. Εστιάζουμε στην υγεία, όχι στην ανάπτυξη. Και όταν λέμε υγεία για την ανάπτυξη, δεν εννοούμε ότι απλώς η υγεία συνεισφέρει στην ανάπτυξη θέλουμε να πούμε ότι αν επενδύουμε στην υγεία, τότε θα αυξήσουμε την ανάπτυξη. Αν οι πολίτες μας είναι υγιείς, αυτό σημαίνει μεγαλύτερη ανταγωνιστικότητα για την Ευρώπη και μεγαλύτερη παραγωγικότητα. Θέλω το πρόγραμμα αυτό για την υγεία να μας απο να δείξει ότι η υγεία δεν είναι ούτε πολυτέλεια, ούτε κοστίζει, αλλά ότι είναι εγγενές τμήμα μιας έξυπνης ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων και εξασφάλιση ενός πανανθρώπινου αγαθού. Θέλω το πρόγραμμα υγείας να επενδύσει περισσότερο στην ε, βιωσιμότητα του συστήματος, ούτω ώστε να υπάρχει καθολικότητα της υγείας και ποιότητα της ποιότητας, ούτω ώστε να μην υπάρξει κανένα συμβιβασμό ε, βραχυπρόθεσμα. Η καινοτομία των συστημάτων υγείας είναι παράγοντες ε, επίτευξης του στόχου της ε, ανάπτυξης. Και αυτό είναι τμήμα της ε, Στρατηγικής Ευρώπη 2020. Αυτό το πρόγραμμα είναι το χρηματοδοτικό μέσο της πολιτικής υγείας. Θα βοηθήσει να εφαρμόσουμε τα εργαλεία για να υλοποιήσουμε την νομοθεσία μας, φερειπίν στην διασυνοριακή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη ή στη φαρμακοεποπτεία. Αυτό το πρόγραμμα δεν είναι ούτε ερευνητικό, ούτε διαρθωτικό πρόγραμμα. Δεν μπορεί να περιμένει κανεί με αυτό το μικρό ποσό να συνεισφέρει άμεσα στην καλύτερη λειτουργία των εθνικών ε, συστημάτων υγεία. Έχει σε σκοπό να εντοπίσει και να δημιουργήσει ε, συνεργασίε και εργαλεία που μπορούν να συνεισφέρουν ε, προ την επίτευξη βιωσιμότητα των συστημάτων υγεία και αντιμετώπιση των ανισοτήτων στον τομέα τη υγεία. Ελπίζω τον Ιούνιο να συζητήσουμε με την Επιτροπή σας αυτό το θέμα. Πάμε τώρα ε, σε σοβαρές απειλές διασυνοριακές για την υγεία. Το Δεκέμβριο πέρυσι η Κομισιόν υιοθέτησε μια πρόταση για να βελτιώσει την ε, ενωσιακή, τον ενωσιακό συντονισμό και την ετοιμότητα ε, για να είμαστε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε τέτοιες απειλές. Βασιζόμαστε σε νέα νομοθεσία για τις μολυσματικές ασθένειες και καλύπτουμε διάφορες απειλές, βιολογικές, χημικές, περιβαλλοντικές ή άγνωστες, ούτως ώστε να έχουμε ένα συνεπές νομικό πλαίσιο για την πρόληψη και τον έλεγχο όλων των κινδύνων. Θέλω να επιληθεί αυτό το σημαντικό ζήτημα, το οποίο είναι φυσικά προς το συμφέρον όλων των Ευρωπαίων πολιτών. Και τώρα πάμε στα τρόφιμα. Και στα εξειδικευμένα μάλιστα τρόφιμα. Οι βασικοί στόχοι της αναθεώρησης που προτείνουμε ε, στους κανόνες στον τομέα αυτό ε, είναι να ενισχύσουμε και να ξεκαθαρίσουμε τις ε, διατάξεις που αφορούν τις ευάλωτες ομάδες πληθυσμού και να προστατεύσουμε τους καταναλωτές από πιθανές, πιθανά προβλήματα λόγω διαφορετικών κανόνων. Θέλουμε μικρότερο γραφειοκρατικό άχθος, περισσότερη συνέπεια και διαφάνεια και μεγαλύτερη ευελιξία για αυτή την ζωντανή και αγορά τροφίμων. Ελπίζω ότι μπορεί να υπάρξει συμφωνία μεταξύ του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου στην πρώτη ανάγνωση. Η Κομισιόν είναι έτοιμη για να παίξει το ρόλο της για να βοηθήσει σε αυτή τη φάση. Μια άλλη σημαντική πρωτοβουλία που τη συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι η πρόταση της Κομισιόν για την καλλιέργεια γαματαφόμικρων, που σκοπό έχει να δώσει στα κράτη-μέλη τη δυνατότητα να μπορούν και αυτά να πούν την άποψή τους για το αν θέλουν ή όχι να επιτρέψουν, αν θέλουν ναι ή όχι να επιτρέψουν την καλλιέργεια γαματαφόμικρων στην επικράτειά τους. Είμαστε σε φάση αποφασιστική και ελπίζω να υπάρξει πολιτική συμφωνία στο Συμβούλιο Περιβάλλοντος τον Ιούνιο. Και τώρα πάμε σε θέματα φαρμάκων. Η Κομισιόν υιοθέτησε το Φεβρουάριο του 2012 ε, χωριστές τροποποιημένες προτάσεις για την ενημέρωση στους ασθενείς και δύο νέες προτάσεις για τη φαρμακοεποπτεία. Οι προτάσεις για τη φαρμακοεποπτεία συμπεριλαμβάνουν διατάξεις για να καλυφθούν τα χάσματα όπως έχουν εντοπιστεί στα τεστ αντοχής ε, που κάνει η Κομισιόν μετά την υπόθεση του Mediator. Ε, Δεδομένη τη σημασία του θέματο, ε, είναι ευπρόσδεκτο το ενδιαφέρον και του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τόσο ώστε να υπάρξει έγκαιρη υιοθέτηση τη πρόταση για τη φάρμακο Αν είναι δυνατόν, πριν τον Ιούλιο που θα τεθεί σε ισχύ η νέα πρόταση για τη φάρμακοεπαγρύπνηση. Θέλω να διδαχθούμε από την υπόθεση του Mediator και να ενισχύσουμε τους κανόνες αυτούς του 2010. Να πάμε παρετέρω από το 2010. Πάμε τώρα ε, στις επόμενες προτάσεις και πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να θέσω το θέμα της αναθεώρησης της οδηγίας για τις κλινικές δοκιμές. Η Κομισιόν σκοπεύει να υιοθετήσει μια πρόταση κανονισμού πριν από τι καλοκαιρινές διακοπέ. Σύντομα, θέλουμε η Ευρώπη να είναι πιο ελκυστική για την κλινική έρευνα. Θέλουμε να αντιστρέψουμε την προβληματική κατάσταση στις κλινικές δοκιμές τα τελευταία χρόνια, χωρίς να δημιουργήσουμε πρόβλημα με τα δικαίωμα των ασθενών, ούτε με την ασφαλειά τους, ούτε να έχουμε πρόβλημα με την αξιοπιστία των δεδομένων. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για την ανάπτυξη νέων φαρμάκων και θεραπείων οι δοκιμέ αυτές όμως συνεισφέρουν και στην ανάπτυξη και σε θέσεις απασχόλησης στον τομέα της δημόσια υγεία, γιατί δημιουργούν σημαντικές επενδύσεις, ελκύουν σημαντικές επενδύσεις. Ελπίζω ότι μπορώ να βασιστώ στην υποστήριξη της Επιτροπής σας κατά τη διάρκεια της νομοθετικής περίοδου για αυτή τη σημαντική πρόταση. Ε, πάμε τώρα στα... στις ιατρικές Θα ξέρετε πολύ καλά ότι η υπόθεση απάτης που έγινε με τα, με τα πρόσθετα στήθους, πώς τα... με τα εμφυτεύματα στήθου, ε, στήθους, ήταν ένα τεράστιο θέμα. Θα παρουσιάσω το συντομότερο δυνατόν για να θεωρήσουμε την νομοθεσία ε, για τα ιατρικά αυτά, τις ιατρικές συσκευές, κάτι που το είχαμε στο μυαλό μας πολύ πριν προκύψει το θέμα με τα εμφυτεύματα στήθους. Θέλουμε να ενισχύσουμε την ασφάλεια των ασθενών και να αποφύγουμε υποθέσεις όπως αυτή με τα εμφυτεύματα. Στο μεταξύ, τα εμφυτεύματα σιλικόνης μάλιστα. Στο μεταξύ, συνεργαζόμαστε με τα κράτη-μέλη <clears throat> για άμεσα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν στο σημερινό κανονιστικό πλαίσιο για να ενισχύσουμε το σύστημα, ιδίω για θέματα που συνδέονται με την εποπτεία τη αγορά και την εποπτεία ε, των φορέων κοινοποίησης. Η Επιτροπή σας ήταν και είναι ε, στεναρός και αποφασιστικός σύμμαχος στον αγώνα κατά του καπνού. Ξέρω ότι το Κοινοβούλιο περιμένει με ανυπομονησία τις επόμενες προτάσεις για την αναθεώρηση της οδηγίας προϊόντων καπνού. Ελπίζουμε στο τελευταίο τρίμηνο του έτους να σας τις κάνουμε αυτές τις προτάσεις. Η πλειοψηφία των ε, καπνιστών ξεκινάει το κάπνισμα ε, στην εφηβεία και μετά δυσκολεύονται να το κόψουν. Από τη σκοπιά της υγείας, ο βασικός μας στόχος θα πρέπει να είναι να μειώσουμε την, το κάπνισμα στους νέους. Θα βασιστούμε σε τρεις βασικούς τομείς. Το πεδίο εφαρμογή, ελκυστικότητα και πρόσβαση. Και μία επιπρόσθετη, ένα επιπρόσθετο στοιχείο θα μπορούσε να καταπολέμηση του παράνομου εμπορίου. Ε, αυτό προέκυψε από την διαβούλευση των ενδιαφερομένων φορέων. Θα θυμάστε, αγαπητοί βουλευτέ, <clears throat> ότι δεν μπορέσαμε να συμφωνήσαμε στην ε, περσινή διαμεσολάβηση επί της πρότασης για τα novel foods ε, με κλωνοποίηση. Η κλωνοποίηση ήταν αυτή που μας διέρεσε. Και τώρα η Κομισιόν αντιμετωπίζει το, την κλωνοποίηση χωριστά από τα υπόλοιπα novel foods ε, και θα κάνει μία χωριστή πρόταση για το, την κλωνοποίηση στις αρχές του 2013. Ε, ελπίζω να έχω την υποστήριξή σας, ούτως ώστε να υιοθετηθούν και οι δύο προτάσεις.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 and to addressing any questions that you may have. Thank you. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Επίτροπε για την ε, εισήγησή τη δήλωσή σας. Έχουμε τώρα 17 συναδέλφους εδώ που έχουν εγγραφεί στον κατάλογο και έχουν ζητήσει το λόγο. Όχι, 19. 19 έχουν ζητήσει το λόγο. κάπνισμα, ιατρικές συσκευές, εργαλεία, ξέρω, όλα αυτά έχουν, θέλουν, αρχίζουν οι συνάδελφοι συντονιστές. Ο κύριος Λίζε ειχε το λόγο για τρία λεπτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε για τη δουλειά σας. Θα ήθελα να αναφερθώ σε δύο μελλοντικά νομοθήματα πρώτα κλινικά πειράματα καλό είναι πως η Κομισιόν κοιτάει το μέλλον, συμφωνούμε με τους στόχους. Θέλω να σας ρωτήσω, να σας ενθαρρύνω, να προχωρήσετε στην καταγραφή των ε, κλινικών πειραμάτων, γιατί δεν δίνονται όλα τα δεδομένα των κλινικών πειραμάτων ε, των ε, φαρμάκων. Εάν δεν είναι θετικά, αποσιωπούνται. Θα μπορούσαμε Όπω σε κράτη, κάποια κράτη-μέλη και στη ΣΥΠΑ, να καταγράφονται τα κλινικά πειράματα. Θα μας βοηθούσε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα που συζητήσαμε πριν από λίγες εβδομάδε στην Επιτροπή, ότι δηλαδή έχουμε κλινικά πειράματα σε τρίτε χώρες μόνο και δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι πως ε, πληρούνται οι προδιαγραφές ε, ποιοτικέ και ηθικές ε, που θέτουμε για τα ευρωπαϊκά γράμμα, φάρμακα. Υπήρχαν ανησυχητικέ πληροφορίε και θεωρώ πω ε, η καταγραφή θα μπορούσε να μα βοηθήσει. Αλλά θέλω να παρακαλέσω την Κομισιόν να δει το θέμα αυτών των πειραμάτων σε τρίτε χώρε. Δεύτερον, αναφέρατε τα ιατρικά προϊόντα και οπωσδήποτε με το ψήφισμα που εγκρίναμε πριν από λίγο ομόφωνα είμαστε στην ίδια γραμμή. Πρέπει να δράσουμε δηλαδή γρήγορα και να έχουμε αναθεωρημένη νομοθεσία. Εάν κατάλαβα καλά, μαζί με τα ιατρικά προϊόντα πρέπει να δούμε και τα διαγνωστικά προϊόντα in vitro. Υπάρχει και σχετική πρόταση. Π.χ. θα ήθελα να αναφέρω ιδιαίτερα το ζήτημα των, των, των τεστ DNA των τεστ ε, DNA ένα διασυνοριακό φαινόμενο. Στέλνει κανείς απλά το αίμα και του στέλνουν τα αποτελέσματα και ό,τι μπορεί να φανταστεί. Χρειαζόμαστε ποιοτικέ προδιαγραφές κατά την άποψη του Κοινοβουλίου γιατί είχαμε γκρίνει ένα ψήφισμα πριν από λίγα χρόνια, χρειάζεται εδώ πέρα μια συμβουλή των ανθρώπων, γιατί έχουν δραματικές επιπτώσεις συχνά στην ζωή των ανθρώπων. Μαθαίνει κανείς ότι έχει γενετική ασθένεια ε, πρέπει να τον βοηθήσουν αυτόν τον άνθρωπο πριν και μετά για να το αντιμετωπίσει σωστά και να γίνει αυτό πριν ε, κάνει το τεστ και όχι αφού πάρει την τρομάρα γιατί αυτό έχει μετά δραματικές συνέπειες. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό και θα ήθελα να το δείτε. Ευχαριστούμε. Λίντα Μακάβαν κατόπιν συντονίστρια των σοσιαλιστών και η για την φάρμακο-επαγρύπνηση που θα συζητήσουμε αύριο πρωί-πρωί. Λίντα. On that item, Commissioner, we are hoping to have... Επίτροπε, ελπίζουμε να συμφωνήσουμε γρήγορα. Τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές, οι συγητές και οι συνεισυγητέ και οι σκιώδες, όλα αυτά να τα τακτοποιήσουμε, να τα Εγώ σήμερα ήρθα σε επαφή με τους υπουργούς, με το Συμβούλιο, ελπίζω όλα να πάνε με το σχέδιο και επομένως θα πρέπει να δούμε αυτά τα, τα, τα, μεγάλα θέματα τα, τα οποία αναφέρατε. Υπάρχει κάτι που δεν μας το είπατε για το ε, Γιώργης, δηλαδή είναι η μεταφορά των ζώων. Όπως ξέρετε έχουμε ε, μια αναφορά με ένα εκατομμύριο υπογραφέ, η ΕΦΣΑ επίσης όπως ξέρετε ε, η Κομισιόν θέλει να, να, να, να αλλάξει τους κανόνες σε σχέση με τις ε, μακρινές μεταφορές και τελικά μετακινήθηκε. Δεν μετακινήθηκε συγγνώμη, η Επιτροπή σε σχέση με αυτό. Αλλά γιατί πιέζει ο χρόνο σα, πιέζει εσά, πιέζει και εμά. Αν επομένω σύντομα δεν προτείνετε κάτι, δεν θα υπάρξει νομοθεσία. Αυτά θέλουν οι Ευρωπαίοι. Ήταν μεγάλη επιτυχία η δουλειά μα όσον αφορά την καλομεταχείριση των ζώων. Επομένω, παρακαλώ, κάντε κάτι όσον αφορά τη μεταφορά. Λίντα, ευχαριστούμε. Επομένω, ο Κρι Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Χαίρομαι που σα ξαναβλέπουμε. Εγώ έχω πονόντο τρομερό σήμερα. Πέστε μας, εσείς, ως Επιτρόπης Υγείας, τι θα κάνει για τον ε, πόνοδοντό μου. Όχι, όχι, όχι. Νομίζω ότι είσαστε πολύ ικανός πολιτικός, αλλά δεν ξέρω αν είσαστε ικανός οδοντίατρος. Τώρα, κάτι πρώτα απ' όλα για τα καλλιντικά. Ξέρετε ότι η σχετική νομοθεσία σε 8 μήνες θα τεθεί σε εφαρμογή και ε, μιλούμε για τα συστατικά των κανονικών που προέρχονται από δοκιμές σε ζώα. Μήπως η Κομισιόν πρόκειται να δημιουργήσει κάποια παραθυράκια, να θεσπίσει κάποιες εξαιρέσεις, ειδικέ περιστάσεις. Δεν ξέρω. Πέστε μας δύο λόγια πάνω σε αυτό, εάν θέλετε να γίνει κάτι τέτοιο. Εάν ισχύει κάτι τέτοιο, θα γίνει με πρωτογενή νομοθεσία ή με κατοξιοδότηση πράξη. μπορούμε να τα συζητήσουμε ούτως ώστε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη περιχαράκωση όσο γίνεται τώρα για τον κύριο συνάδελφο Μάντερς ο οποίος πρέπει να φύγει σε λίγο είχε επισημάνει η Κομισιόν σχετικά με τους κινδύνους από τα τρόφιμα τι λέτε εσείς ε, γιατί έχετε θέματα για καταναλωτές Τι θα κάνει η Επιτροπή όσον αφορά κάποιου είδου πρωτοβουλίε για αυτό το θέμα των τροφίμων. Thank you very much, Chris. Now for the Greens, Michel Ivazi. Μισελ, για τους πράσινους. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας κύριε Επίτροπε. Εγώ έχω πάρα πολύ συγκεκριμένη ερώτηση. Και αυτό γιατί μας πλησίασαν και απευθύνθηκαν σε εμάς η μη κυβέρνηση οργανώσει για τα λοιπά μα είπε ότι οι φυτογενικέ υπηρεσίε έχουν μέχρι το 2008 και το 2012 για να διδύσουν την αγορά ένα σωρό τέτοια, τέτοια ε, τα οποία όμω θα τα αποσύρουν μετά. Δηλαδή οι επιχειρήσει αποσύρουν τα προϊόντα του γιατί δεν τηρούνται υγειονομικέ διατάξει για το περιβάλλον. Όμω μπορούν ε, ε, ε, σύμφωνα με έναν κανονισμό των 33 του 2008 του Ιανουαρίου του 8 να ξαναρίξουν στην αγορά αυτά τα ε, με κάποια διαδικασία που λέγεται επανυποβολή. Επομένως, αυτό είναι κάτι το οποίο μας απασχολεί πάρα πολύ, γιατί υπάρχουν ένα σωρό επιστήμονες, Γάλλοι και Βρετανοί, οι οποίοι πρόσφατα στο περιοδικό Science λέει ότι τα νοικοτινοειδή είναι κάποια συστημικά φάρμακα τα οποία σκοτώνουν τις, ε, τις, τις, τις μέλισσες ε, και, και, άλλα έντομα. Επομένως, υπάρχει μεγάλος κίνδυνος για την υγεία. Πεςτε μας, εσείς τι λέτε. Πρόκειται περί ευρωπαϊκού κανονισμού. Έχουμε την οδηγία του 99, 91, συγγνώμη, του που, που, που θεσπίζει αυτή την εξαίρεση για αυτά τα προϊόντα με τα οποία δημιουργούν αυτό το μεγάλο κίνδυνο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο τελευταίο ομιλητή για τι πολιτικέ ομάδε είναι η κυρία Λιωτάρ. Ευχαριστώ, ευχαριστούμε κύριε Ντάλη που ήρθατε εδώ πέρα για να ανταλλάξουμε απόψεις. Χάρηκα που είπατε πως θα καταθέσετε δύο διαφορετικές προτάσεις. Μία για τα καινοτόμα τρόφιμα και μία για την κλωνοποίηση. Η κλωνοποίηση μας απασχολεί όλο και περισσότερο. Και θέλω να σας ρωτήσω, ξέρετε τι ή ποιος είναι το πανκ πανκ. <laughs> Ναι, σας βλέπω έτσι που κοιτάτε με απορία. Για τους συναδέλφους που δεν ξέρουν, να εξηγήσω. Χτες στις ειδήσει είδαμε πως υπάρχει ένα, στην Κίνα ένα νέο πρόβατο που ονομάζεται Bang Bang. Ε, Διασταύρωση μεταξύ προβάτου γενετικώς τροποποιημένου και μετά κλωνοποιημένου για να έχει καλύτερη απόδοση το οποίο μετά όμως προσβλήθηκε από ταινία του στομάχου ένα σκολικό πρόβατο δηλαδή Δηλαδή ξεκίνησαν να φτιάξουν ένα καλό διατροφικό προϊόν που θα είχε θετικά λύπη υποτίθεται, αλλά το αποτέλεσμα ήταν αυτό το ολέθριο. Εν ολίγης, μπορούμε να απαγορεύσουμε τέτοια τρόφιμα ή πρέπει να κινηθούμε ακόμη πιο γρήγορα με την ομοθεσία μας. Δεύτερον, σε σχέση με αυτό το οποίο είπε η Λίντα Μακάβεν για την μεταφορά των ζώων, ξέρουμε πως η πλειοψηφία α, του Κοινοβουλίου είχε απευθυνθεί στον εκπρόσωπό σας για το ότι δεν προβλέπεται αναθεώρηση του κανονισμού υπαριθμών 1 του 2005 για τη μεταφορά των ζώων και είχατε πει πως πρόκειται περί παρεξήγησης και πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη μεταφορά των ζώων και άλλη μια ερώτηση για την ασφάλεια των τροφίμων την πρόταση σας για το διατροφικό προφίλ πότε μπορούμε να την περιμένουμε Ευχαριστούμε πολύ. Τώρα τέλειωσε ο πρώτο γύρο. Έχουμε τώρα ένα σώρο ερωτήσει. Ακόμα και για το πανκ πανκ έχουν υποβληθεί ερωτήσεις για την καλομεταχείριση των ζώων. Και τώρα παρακαλώ ο κύριος Επίτροπος αν θέλει μπορεί να απαντήσει αυτές τις ερωτήσεις. Κύριε Νταλή έχετε το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ λέει ο Επίτροπος. Ας αρχίσουμε με τον Πίτερ, Πίτερ Λίζε και τις ε, κλινικές δοκιμές. Ναι, λαμβάνονται υπόψη αυτά τα οποία είπατε για τις νέες μας προτάσεις τις οποίες και θα υποβάλλουμε. Πάντως, αυτό το οποίο θέλουμε να κάνουμε είναι τώρα οποιαδήποτε κλινική δοκιμή η οποία καλύπτεται από αυτήν την διαδικασία έγκρισης θα πρέπει να έχει προαναγγελθεί πριν ξεκινήσει και να έχει γίνει σχετική κοινοποίηση. Ακόμα και αν λαμβάνει χώρα εκτός Ευρώπης. Αυτό αποσκοπεί στο να ελέγχονται οι κλινικές δοκιμές και να εξασφαλίζεται ότι τα κριτήρια τα οποία χρησιμοποιούνται είναι τα ορθά και ότι μας ενημερώνεται για οποιοδήποτε αποτέλεσμα αυτών των δοκιμών. Διότι ακόμα και τα αρνητικά αποτελέσματα βοηθούν την επιστήμη. Οπότε και οι επιστήμονες λοιπόν είναι σημαντικό να ενημερώνονται για το τι γίνεται. Τώρα όσον αφορά για το DNA, για τα άλλα τεστ in vitro, κατανοώ τα θέματα που αναγκύπτουν είναι κυρίως ηθικής φύσεως θέματα κρατών μελών. Για την φαρμακοεπαγρύπνηση, α, με χαρά μου, μαθαίνω ότι όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο. Και πρόσφατα άκουσα ότι είχαμε κάποιες διαταράξεις από πλευράς Συμβουλίου, αλλά τα πράγματα εξομαλύνθηκαν. Οπότε για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό, διότι νομίζω ότι έχουμε συγκεκριμένες απαντήσεις. Πρόκειψε σαφώς ότι θα πρέπει οι διαδικασίες ε, αναφοράς, έκθεσης να διέπονται από αυτές δύο τάξεις. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα εγκριθούν τελικά. Τώρα όσον τη μεταφορά των ζώων. Και σε σχέση και με αυτό που είπε η κυρία Λεωτάρ. Έχουμε λάβει υπόψη το θέμα. Και η θέση μας είναι ότι ισχύει τώρα κανονισμός που αφορά τη μεταφορά των ζώων. Και δυστυχώ ξέρουμε ότι η εφαρμογή αυτού του κανονισμού δεν είναι στα επίπεδα τα επιθυμητά. Οπότε και εμείς θα πρέπει πρώτα-πρώτα να επιμείνουμε, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι αυτές οι διατάξεις εφαρμόζονται χρησιμοποιώντας σύγχρονα μέσα τεχνολογικά για την εφαρμογή. Τα έχουμε. Τώρα για το κατά πόσο εγώ συμφωνώ ότι θα πρέπει να είναι όσο γίνεται συντομότερη αυτή η διαδρομή, Απλώς σας εγώ αυτό που έχω πει δημοσία, επανειλημμένως πιστεύω, ότι θα πρέπει να, να περιορίζονται στο, στο ελάχιστο δυνατό αυτές οι μεταφορές. Και όπως οι περισσότεροι εξημών γνωρίζετε, Οπότε, Υπάρχει σχετική θέσια που λέει πού σφάζεται το ζώο, από πού ξεκινάει, πού μεγάλωσε. Άρα θα πρέπει στην πηγή να αντιμετωπίζετε το θέμα. Τι δηλαδή, από πού ξεκινάει, τι προκαλεί ούτω ή τη μεταφορά. Αυτή είναι η άποψή μου. Πριν επομένω ξεκινήσουμε όλα τα, τα, τα, τα, τα, περίπλοκα μέτρα για για τη μεταφορά, για τα σχετικά. Γιατί έχουμε μεταφορά των ζώων. Τα ρουμανικά άλογα λένε ότι είναι Ιταλικά στην ετικέτα γιατί τα σφάζουν στην Ιταλία όταν έχουν ε, ανατραφεί, όταν έχουν εκτραφεί μάλλον στην Ρουμανία. Ε, το, το, προϊόν είναι ρουμανικό και όχι ιταλικό. Ένα απλό παράδειγμα είναι αυτό. Αυτά πρεσβεύω. Σας λέω την αλήθεια. Και επομένως ποντάρω στη δική σας συνεργασία, ούτως ώστε να αποσπάσουμε κάποιο αποτέλεσμα, κάποια λύση όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων. Όσον αφορά τα καλλιντικά. Τα θέματα τα οποία έχουμε αφορούν το ότι παρά το ότι έχει σημειωθεί πρόοδος από τη βιομηχανία των καλλιντικών και αυτό αφορά και είναι αποτέλεσμα και της νομοθεσίας που έχετε θεσπίσει εσείς, έχουμε αντικαταστήσει αυτά, τα, αυτές τις δοκιμές με εναλλακτικού τρόπους δοκιμών. Πολύ καλό. Έχει επενδυθεί πολλά και παρόλα αυτά όμως για κάποιε περιπτώσει ακόμα δεν έχουμε εναλλακτικέ λύσει. Όταν επομένω, ζήτησαν να μου πούν Τι χρονοδιάγραμμα υπάρχει για να εξευρεθεί η λύση. Αναφέρθηκε, μου απάντησαν για κάποια εξαετία, αλλά και για κάποιες άλλες δοκιμές είπαν ότι ακόμα δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς πότε θα έχουμε ελεκτική. Αφού επομένω δεν έχουμε κάποιο, κάποιο, κάποια προθεσμία, κάποια ημερομηνία για το πότε μπορούμε να έχουμε μεθόδους ελεκτικές, τότε αναβάλλεται η θέσπιση της σχετικής νομοθεσίας. Σαν να αναβάλουμε μόνος λήψη απόφαση. Μου φαίνεται λογικό να πούμε ότι η νομοθεσία θα πρέπει να θεσπιστεί όπως προβλέπεται, όπως προγραμματίστηκε. Άρα τελικά να μην υπάρχει καμία αναβολή. Από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι θα πρέπει να επιτρέψουμε κάποια δυνατότητα για κάποια προϊόντα καινοτόμα, κάποια συστατικά που να συνεχίσουν να παράγονται. Και θα προτείνουμε σύστημα νέων παρεκκλήσεων, ούτως ώστε οι Ευρωπαίοι να μπορούν να έχουν πρόσβαση σε νέα προϊόντα καλλιντικών και να μπορεί η βιομηχανία να, να λέει στην ότι αυτά έχουν παραχθεί κατόπιν δοκιμών σε ζώα. Θα πρόκειται για συγκεκριμένες παρεκκλήσεις. Και αυτό θα περιχαραγώνεται από πολύ αυστηρές διατάξεις. Επίσης, έχει ζητηθεί πιο ευελικτή ερμηνεία, ούτως ώστε να μπορεί η βιομηχανία να χρησιμοποιήσει κάποια δεδομένα τα οποία ε, προέρχονται και εκτός και, και, και, και από τρίτες χώρες, ούτως ώστε αυτό να αφορά και άλλα προϊόντα εκτός από τα ελληνικά, όπως για την φαρμακευτική έρευνα βάσει του REACH. Ό,τι αλλαγή και να γίνει, Κύριε Βάνη, θα, θα, θα, γίνεται με πρωτογενέ δίκαιο, τέτοιε διατάξει πρωτογενή νομοθεσία και θα είναι επομένω αυτό μια ευκαιρία, ούτω ώστε να υπάρχει 100% εποπτεία έλεγχο και όπω είπατε και εσεί σωστά, θα μπορέσουμε έτσι να, να αναχτενίσουμε αποτελεσματικά τι νέε διατάξει. Τώρα, όσον αφορά τα απόβλητα, τα απορρίμματα που προέρχονται από είδη διατροφής. Ο συνάδελφος Ποτόσνικ ε, ασχολείται με αυτό, αλλά πάντως έτσι κι συνεργαζόμαστε πολύ με τον Ποτόσνικ και τις υπηρεσίες του. Και περί τα τέλη του έτους θα έχουμε μία πρόταση για την βιώσιμη κατανάλωση και κάποιο κοινό συμπόσιο, κοινή διάσκεψη θα οργανώσουμε. Ούτω ώστε να είναι υψηλή προτεραιότητα σε κάθε μας δράση. Είναι θέμα περιβάλλοντος πρώτα-πρώτα, αλλά είναι και θέμα ε, της ε, βιώσιμης φύσης των, των τροφίμων. Και είναι και θέμα της οικονομικής πραγματικότητας. Το πώς θα εκπαιδεύσουμε τους Ευρωπαίους ούτως ώστε να μπορούν να διαχειριστούν το το του τροφίμων τους καλύτερα. Βέβαια το θέμα είναι ευρύτατο. Το θέμα δεν είναι μόνο το τι αγοράζουν οι Ευρωπαίοι, αλλά και πώς προσθέτει το προϊόν, η συσκευασία, ας πούμε. Αν τελικά το μισό αυτό που αγοράζουν το πετάνε. Μας απασχολεί επομένως αυτό πολύ. Τώρα τα ζενιοκτώνα, τα φυτοφάρμακα. Το 2009 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θέσπισε ένα νέο νομοθετικό πλαίσιο. Έναν κανονισμό. Οπότε και εμείς σε συνέπεια αυτού θα πρέπει να επανεξετάσουμε το θέμα τι φάρμακα κυκλοφορούν δηλαδή στην αγορά, τα οποία ήδη είχαν αυτήν την ρήτρα sunset. Σταδιακής λήξης. Πάντως τώρα έχουμε θεσπίσει ένα χρονοδιάγραμμα. Ένα χρονικό πλαίσιο, βάσει το οποίο θα γίνει κάποια αναθεώρηση ε, σύμφωνα με την κοινωνική νομοθεσία για ε, τις διατάξεις που αφορούν αυτά τα φάρμακα. Για τώρα για το πανκ-πανκ και την κλωνοποίηση. Όπως είπε η κυρία και η κυρία Λιωτάρ, το συζητήσαμε, το συζητήσαμε τότε σε εκείνη την ε, διάσκεψη με τις ώρες. ή Υπόσχεθήκαμε να κάνουμε μία αξιολόγηση επιπτώσεων για την κλωνοποίηση συνολικά, την ετικετοθεσία κλπ. Όλα τα θέματα που ανέκυψαν πρόκειται να καλύπτονται από αυτήν την μελέτη των επιπτώσεων. Άρχισε αυτό που υποσχεθήκαμε. Μην το βραχυκλώνουμε. Ε, ε, μην, μην, μην βραχυκλώνουμε ούτε την αξιολόγηση αυτή, ούτε τη σχετική μελέτη. Άρα, αρχάς το 2013 θα προκύψουν τα αποτελέσματα τα οποία βεβαίω και θα σας υποβάλουμε στη συνέχεια για την κλωνοποίηση, οπότε μετά μπορούμε να συζητήσουμε για νομοθεσία ειδικότερη για την κλωνοποίηση, ακριβώ, όπως έχουμε υποσχεθεί ότι θα πράξουμε. Αυτό το οποίο εγώ θέλω να δω είναι, στο μεταξύ χωρίς να περιμένουμε, για αυτές τις ενέργειες, για, το, για την κλωνοποίηση, να προχωρήσουμε στο θέμα των ειδών διατροφής και αυτό που είπατε και εσείς να γίνει, για που δεν έχουν την κλωνοποίηση να γίνει μια αναθεώρηση ούτω ώστε σύντομα και ταχαίως για τα νέα τρόφιμα να έχουμε κάτι. Να έχουμε όμως μια παραγράφο που να περιορίζει το θέμα της κλωνοποίησης χωρίς όλες αυτές τις λεπτομέρειες. Οπότε και γι' αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ένα νομοθέτημα. ούτως ώστε να μπορούμε να ελέγξουμε και το πανκ πανκ και άλλα προϊόντα. Αυτό προτείνω. Περιμένω όμως από εσά να μου δώσετε το πράσινο φως. Να προχωρήσουμε έτσι με το fast track μια οδηγία για τα νέα είδη διατροφής και κάποιους περιορισμούς για την κλωνοποίηση και να περιμένουμε για μια, μια ένα άλλο νομοθέτημα ευρύτερο για την κλωνοποίηση. και μετά την αξιολόγηση των επιπτώσεων συνεχίζουμε όταν θα έχουμε τη σχετική πρόταση. Όμως, περιμένω εσείς να μου δώσετε το πράσινο φως και να μου πείτε πώς θα πούμε να κινηθούμε. Όσον αφορά τώρα το προφίλ διατροφής. Ή τα προφίλ διατροφής, γιατί συνεχίζουμε τη μελέτη. για αυτά τα θρεπτικά συστατικά. Είναι δύσκολο το έργο μας, αλλά θα το χειριστούμε όσο καλύτερα γίνεται. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε για τις ε, χρήσιμες ε, και πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Ε, αυτό το θέμα Τη μείωση των καταλήπων των τροφίμων είναι παγκόσμιο πρόβλημα. Και ξέρω ότι ο κύριος Ποτόσνικ ασχολείται με αυτό το θέμα, ώστε να υπάρξουν τα αποτελέσματα. Πάμε τώρα στο δεύτερο γύρο με 14 βουλευτές. Θέλω να δώσω και στους 14 την δυνατότητα να κάνουν ερωτήσεις. Αυτό σημαίνει όμως ότι θα πρέπει να περιοριστούμε όλοι σε 1,5 λεπτό, ούτω ώστε να μπορέσει να απαντήσει και ο Επίτροπος. Η κυρία Γκοστέτ πρώτη. Κρίμα είναι που μου δίνετε μόνο 1,5 λεπτό γιατί θέλω να πω πολλά. Είμαι εισηγήτρια για το πρόγραμμα υγείας. Θέλω καταρχάς, Επίτροπε, να σας συγχαρώ γιατί στην Επιτροπή ε, επιτύχατε το 5,7% αύξηση των προγραμμάτων υγείας σε σχέση με το τι είχαμε μέχρι τώρα. Σε περίοδο κρίσης αυτό είναι επίτευγμα. Μπράβο, θα σας υποστηρίξουμε. Ε, έχω μια μικρή διαφωνία, όπως ξέρετε, όμως, για τον τίτλο. Ο τίτλος σας είναι ε, «Υγεία για την ανάπτυξη». Εγώ θα προτιμούσα «Υγεία και ανάπτυξη», γιατί θεωρώ ότι η υγεία δεν εξυπηρετεί μόνο την ανάπτυξη. Τέλος πάντων, το συζητήσαμε αυτό και νομίζω ότι θα το συζητήσει και η Επιτροπή αυτό το θέμα. Οπότε το προσπερνάω γρήγορα. Θέλουμε η δημοσιονομική κατανομή ανάμεσα στους τέσσερις στόχους του προγράμματος, ενίσχυση της κοινότητας, βελτίωση στην πρόσβαση των ε, ε, ε, υπηρεσιών υγείας, να προστατεύσουμε τους πολίτες από τις απειλές, όλα αυτά να μην είναι στατικά για να μπορεί το πρόγραμμα αυτό να παρεμβαίνει όταν υπάρχει ανάγκη. Επίση, πρέπει να σκεφτείτε και τι συνέπειε τη γύρα του πληθυσμού. Επομένω, πρέπει να το δούμε μαζί σα το θέμα αυτό, Επίτροπε, και με την Δανέζικη Προεδρία. Γρήγορα, το δεύτερο θέμα. Ε, τα Ιαπωνέζικα προϊόντα καταλαμβάνουν και περισσότερο μερίδιο τη αγορά. Ε, Μα ανησυχεί όμω σε επίπεδο υγεία, γιατί υπάρχουν πάρα πολλά βακτηρίδια μέσα σε αυτά. 51% των κινέζικων προϊόντων ε, αποτυγχάνουν στου ελέγχου. Όμω, έχουμε το γάλα με τη μελανίνη, ε, Έχουμε ε, τόφου που έχουν πρόβλημα, έχουμε ζελατίνη ε, στα, στις γαρίδες. Όλα αυτά είναι πολλά, πολύ προβληματικά, πολύ σοβαρά. Επίσης τα εδάφη στα οποία καλλιεργούνται στην Κίνα είναι μολυσμένες από βαρέα μέταλλα. Όλοι το ξέρουν. Εσείς θεωρήσατε ότι η Κίνα δεν είναι αρκετά ασφαλής χώρα. Θα θέλαμε να μας δώσετε κάποια στοιχεία για αυτό το θέμα, γιατί μου φαίνεται πάρα πολύ σοβαρό. Συνεχίζουμε. Ευχαριστώ που ήρθατε στην Επιτροπή μας, κύριε Νταλή. Συμφωνώ ότι ε, υγεία και ανάπτυξη θα, είναι, θα πρέπει να είναι ο τίτλος και όχι η υγεία για την ανάπτυξη. Ε, Επίση, ε, πρέπει να δώσουμε μεγάλη σημασία στην πρόληψη. Ε, χαίρομαι ότι πριν το καλοκαίρι θα έχουμε το θέμα των κλινικών δοκιμών. Κάτι πρέπει να μα δώσετε. Μέχρι στιγμή δεν πάει καλά το, το θέμα αυτό. Κάτι πρέπει να μα πείτε λοιπόν. Το βασικό μου θέμα όμω είναι ε, τα πρώτα καπνού. Ε, με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό. Το θέμα το ξέρετε είναι από τα πιο σημαντικά νομοθετήματα αυτής της Επιτροπής μας. Ε, ξέρετε ότι ο καπνός δημιουργεί πρόβλημα στη δημόσια υγεία, επιβαρύνει τα συστήματα υγεία κτλ. Προσπαθείτε να έχουν γίνει πάρα πολλά για να καταπολεμήσουμε τον καπνό, το ξέρω. Αλλά είναι κρίμα που περιμένουμε το τέλο του 2012 για τι προτάσει, αλλά να τι είχαμε τι προτάσεις ήδη. Περιμέναμε ήδη πάρα πολύ. Ελπίζουμε να κινηθείτε πιο γρήγορα. Δεν είναι σωστό να μας δώσετε μόνο στο τέλο του 2012. Ελπίζω να μην μα καθυστερήσετε κι άλλο. Ελπίζω επίση να υπάρξουν σκληρά μέτρα από εσά στι προτάσει σα για να αντιμετωπίσουμε τον καπνό. Ξέρω ότι υπάρχει φοβερό λόμπινγκ από την ε, καπνοβιομηχανία. Ένα από τα θέματα που λένε είναι το πρόβλημα του παράνομου εμπορίου. Το θέμα τη συσκευασία. Ελπίζω να κάνουμε κάτι. Γιατί ε, νομίζω ότι είναι στην πραγματικότητα μια δικαιολογία. μα παραπλανά αυτό το επιχείρημα. Ε, κάτι θα πρέπει να μα πείτε για το θέμα τη συσκευασία λοιπόν. Και ελπίζω να συνεργαστούμε το συντομότερο δυνατόν. Είναι πολύ σημαντικό για τον κόσμο. Ε, δεν μπορούμε να καθυστερούμε άλλο. Ευχαριστώ, Γκλένις, Σνέλχαρντ και μετά Γιολάινεν. Ευχαριστώ, κύριε Επιτρόπε, που ήρθατε τώρα για το εάν θα πρέπει να έρθει πιο νωρίς ο κανονισμός για τα νέα τρόφιμα. Ναι, γιατί έχουμε τόσα πολλά νέα τρόφιμα. Αυτή είναι η δική μου απόψη, δεν ξέρω εάν συμφωνεί ολόκληρη η Επιτροπή. Τώρα, εμείς περνάμε νόμους εδώ πέρα και δεν του εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη. Και διαπιστώνουμε συνεχώς πως πάρα πολλά κράτη-μέλη δεν το κάνουν αυτό. Υπάρχουν σοβαροί λόγοι για αυτό ή όχι. Και θα τιμωρήσετε κάποιε χώρε για να γίνει τίποτα και να εφαρμοστούν οι νόμοι που ψηφίζουμε. Δεύτερο ερώτημα. Αντίσταση στα αντιβιωτικά, κάτι το οποίο μας απασχολεί. σκοπεύεται να υπάρξει ένα μέτρο που θα ισορροπεί και, στον, ε, και θα ισχύει και για τους ανθρώπους και για τα ζώα ή τι προγραμματίζεται ακριβώς ε, τι θα γίνει επίσης γιατί από ό,τι φαίνεται τα μέτρα θα ε, περάσει πάρα πολύ καιρό μέχρι να υιοθετηθούν Επίσης, ε, όσον αφορά τα φάρμακα των ζώων πρέπει να γίνει κάτι. Επίσης, να αναφέρω τα πάρα πολύ αυτά προγράμματα τα οποία αναφέρατε για την ε, υγεία, τα οποία κάνουν καλή εντύπωση στα κράτη-μέλη και νομίζω πως μπορούμε πράγματι να διαφημίζουμε έτσι την Ευρωπαία. Αν συνεχίσετε να κάνετε τέτοια προγράμματα, πραγματικά θα μας ικανοποιήσετε. Μάλιστα, Γιώλα Λάινεν και μετά η κυρία Λεπάζ. Ναι, κύριε Επίτροπε. Σας ε, καλωσορίζουμε τώρα. Η πρόταση αυτή την οποία αναφέρατε δεν έχει πολύ νόημα το σύνθημα αυτό το Health for Growth το Health for Growth δεν βγαίνει στις άλλες γλώσσες κάτι άλλο πρέπει να βρείτε το σύνθημα τώρα για την νομοθεσία για τα νέα τρόφιμα. Συμφωνούμε όλοι εδώ πέρα, πρέπει να την περάσετε. Δεν γίνεται αλλιώ. Και μα έχει υποσχεθεί πω το 2013 θα έχουμε νομοθεσία για την κλωνοποίηση. Νομίζω πω και ο νέο πρόεδρο, ο Ματία, πρέπει να σα δώσει ένα μήνυμα. Η πλειοψηφία των συντονιστών θεωρούσε πω πρέπει να γίνει αυτό. Και έτσι πρέπει να γίνει άρα. Τρίτον, έβδομο πρόγραμμα πλαίσιο, είμαι ο εισηγητής, έχουμε ένα ολόκληρο κεφάλαιο για το περιβάλλον και την υγεία και η Ολομέλεια την Παρασκευή που μας πέρασε ζήτησε ένα δεύτερο πρόγραμμα. Γιατί το προηγούμενο είναι από το 2004, δεν ξέρω αν ε, είναι δικό σας θέμα ή συναδέλφου σας, γιατί υπάρχουν διάφορες σχέσεις μεταξύ υγείας και περιβάλλοντος. Τέλος, ε, καρκίνος του δέρματος Έρχομαι από ένα μεγάλο συνέδριο με τον Αλόης Πέτερλε και λοιπούς της, στην Κοπενχάγη. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ένας κανονισμός πως κάτω από τα 18 χρόνια απαγορεύεται να πάει κανείς στο σολάριουμ γιατί αποδεδειγμένα προκαλούν τα σολάριουμ καρκίνο του δέρματος. Πρέπει να κινητοποιηθείτε. Είναι ένα πρόβλημα που αυξάνεται και ο πληθυσμός της Ευρώπης βεβαίως γυράσκει και θα έχουμε όλο περισσότερες τέτοιες περιπτώσεις. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές Κάτι πρέπει να μας πείτε γι' αυτό. Ευχαριστώ. Κορίν Λεπάζ, είναι... η Κορίν Λεπάζ δεν είναι εδώ. Κυρία Evans. Thank ευχαριστώ Πρόεδρε και ευχαριστώ και τον κύριο Επίτροπο. Μας είπατε ότι περιμένετε να προκύψει τον Ιούνιο στο Συμβούλιο Συμφωνία για ε, τους γενετικά τρομμένους οργανισμούς. Τι γίνεται με τις ε, εισαγωγές διαφόρων τροφών για ζώα και για ανθρώπους που δεν είναι εγκεκριμένα και ε, περιμένουμε να βγάλετε και κάποια μέτρα και για τους σπόρους. Γιατί πάντως όλη την Ευρώπη ξαπλούν τέτοια προϊόντα. προσοχή γιατί και ο κόσμος αλλά και το κοινοβούλιο θα ήθελε να προσέχετε περισσότερο τους γάμματα φόμικρον. Ο τελευταίος ομιλητής τώρα. Κυρία Γιούσο. Και, και κατόπιν και η κυρία Καλνούμπα. Σα ευχαριστούμε για όσα είπατε, κύριε Επίτροπε. Συμφωνούμε 100% σε όσα είπατε για την φαρμακοπαγρύπνηση. Καλά τα είπε και η κυρία Έβανε. Αλλά όσον αφορά την ε, καλομηγία των ζώων εγώ χαίρομαι πάρα πολύ το, το ότι απολαμβάνουν, απολάβουν τέτοιες ε, Εμεί Εμείς, από την άλλη μεριά, ταξιδεύουμε στο αεροπλάνο και είμαστε στριμωγμένοι, σαν σαρδέλες. Είπαμε ότι έχουμε τον εκατομμύριο υπόγραφες, αλλά τι θα γίνει. Άρα, θα γίνει κάτι όπως είπαμε και για τα ζώα και για τους ανθρώπους στα, στα αεροπλάνα και να, να, να, να απομακρυνθούν κάπως τα καθίσματα μεταξύ τους. Τώρα, το θέμα δεν είναι επομένω να μαζεύουμε υπογραφέ, αλλά να μαζεύουμε επιστημονικέ εκθέσει από τη ΕΦΣΑ. Και τι λέει ΕΦΣΑ. Δεν είναι θέμα ορών διαδρομή, αλλά συνθήκων διαδρομή μεταφορά. Εδώ πέρα, για τη κλωμδιακή των ζώων, έχουν πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα. Αυτά όλα θα πρέπει να τεθούν τραπέζι για όλα τα ζώα και τα ζώα τα οποία έχουν σφαγεί. Γιατί ξέρετε, δεν θα πρέπει να έχουμε δύο σφαγή ας πούμε σε πιο κοντά από 10 χιλιόμετρα γιατί είναι τόσο αυστηρές οι προϋποθέσεις που τάσσονται που είναι, είναι οικονομικά. Έτσι κόνουν και τιμές. Πάντως εισάγουμε ζώα για άλλα προϊόντα διατροφής ζωικά από χώρες που δεν έχουν τέτοιους περιορισμούς. Άρα, ή θα παγκοσμιοποιηθούμε ή τίποτα. Να τα αυγά που τρώμε. Είναι ε, προέρχονται από, από, από, από, από κότες που είναι σε κλουδιά 350 τετραγωνικών ενώ τα, οι δικές μας ε, οι δικές μας είναι σε κλουβιά διπλάσια. Θα πρέπει, πρέπει να είναι σε κλουβιά 700 τετραγωνικών εκατοστών. Η τελευταία αλλά σημαντική κυρία Κάλτενμπαχ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τον κύριο Επίτροπο ε, για το ότι έρχεται τόσο συχνά εδώ πέρα. Θέλω να αναφέρω κάποια σημεία. Ήδη αναφέρθηκε η οδηγία την οποία αναμένουμε από εσά το δεύτερο εξάμεινο του έτους. Σας παρακαλέσω να δείτε τις ουσίες οι οποίες προκαλούν ε, εξάρτηση και είναι δηλητηριώδεις ε, εντός αυτής της οδηγίας και να τις απαγορεύσετε. Δεύτερον, ε, θέλω να συμφωνήσω με τον κύριο Λάινεν εδώ πέρα. Το όνομα που έχετε επιλέξει δεν είναι σωστό. Εγώ θεωρώ πως πρέπει να πείτε health literacy Θα πρέπει δηλαδή να μπορούν να βρουν την πρόσβαση μόνοι του στο σύστημα υγείας οι πολίτες της Ευρώπης. Και τρίτον, αυτό το οποίο σα ζητάτε, να ε, θέσετε αυτά τα θέματα στην κοινή γεωργική πολιτική, γιατί πολλά από τα προβλήματα που αντιμετωπίζουμε προέρχονται από μια γεωργική πολιτική που δεν πάει στη σωστή κατεύθυνση. Και ζητάω εδώ πέρα τη στήριξή σα γι' αυτό. Σα ευχαριστώ. Να σας πω πως... Ε, μην ξεχνάτε πως ε, στα γερμανικά λέγεται Öffentliche Gesundheit αντί για Volksgesundheit και τα δύο σημαίνουν βεβαίω δημόσια υγεία στα ελληνικά. Απλά ήταν ο ένα όρο φορτισμένο για ιστορικού λόγου. Κύριε Επίτροπε, λοιπόν, έχετε τον λόγο. Ναι, είναι αλήθεια ότι τώρα υπάρχει αυτό το θέμα για τον τίτλο του προγράμματο και γι' αυτό και ελπίζω όμω ότι πέρα το τίτλου και η ουσία και η ουσία θα είναι καλύτερη και θα είναι πιο αποδεκτή. Όχι, δεν πρόκειται να τσακωθούμε για τον τίτλο, όμως, όμως θα πρέπει να καταλήξουμε σε έναν εύστοχο τίτλο. Health και ανάπτυξη, υγεία και ανάπτυξη, health and growth. Ε, εξίσου αντιμετωπίζονται από το πρόγραμμα. Όχι, δεν μου αρέσει αυτό. Όχι, δεν θα πρέπει στην ίδια ζυγαριά να τα βάζουμε όταν έχουμε ένα πρόγραμμα για την υγεία και να λέμε ότι η ανάπτυξη είναι μια πλευρά της ε, υγείας κλπ. Βέβαια, φυσικά. Ε, εγώ πιστεύω και ήδη έχω μιλήσει με την κυρία Κροστέτ γι' αυτό. Θα πρέπει να κάτσουμε και να στύψουμε το μυαλό μας και να βρούμε μία σύντομη περιγραφή που να ε, αντικατοπτρίζει το πρόγραμμα το περιεχόμενο πρόγραμμα δηλαδή. Και γιατί θέλουμε έτσι να παρουσιάσουμε το θέμα ανάπτυξης; ανάπτυξη. Ε, και, εκεί το βλέπετε, θα σας τα λέω ευθέω. Αναφέρουμε την ανάπτυξη γιατί η ανάπτυξη έχει γίνει το, το, το, το, το, το, πάγιο σύνθημα. Ε, έχει γίνει το, το, το κλειδί για κάθε μεσομικό θέμα. Όχι, δεν μου αρέσει να, να, να, να μιλάω για τα οικονομικά της υγείας. Όμως, όμως είμαστε πολιτικοί. Είμαστε πραγματιστές, ρεαλιστές και ξέρω ότι για, να ανοίξει ο Κορβανάς το χρηματοκιβώτιο το οποίο θα, θα μας χρηματοδοτήσει θα πρέπει να μας καρεύουμε, να, να, να φτιασιδώνουμε έτσι το πρόγραμμα. Να το, να, να, το, να, το, να το περιβάλλουμε, να το στολίζουμε με την οικονομική αργό. Και έτσι να μπορούσαμε να πετύχουμε το τελικό μας στόχο του να πετύχουμε το να έχουν υγεία οι πολίτες μας. Όλοι οι Ευρωπαίοι. Πλούσιοι και φτωχοί. Όπου και να βρίσκονται. Από οποιαδήποτε εθνοτική ομάδα προέρχονται, αυτός ο στόχος μας και επίσης να είναι τα συστήματα υγείας βιώσιμα, αηφόρα. Αυτό, αυτό, αυτό, αυτό με μετρώει και με προβληματίζει. Σας το ομολογώ. Ήδη στη Δανία το παραδέχθηκα ενώπιον των αρμοδίων του Υπουργού Υγείας προσοχή μην βρεθούν αυτοί στο τιμόνι της Ευρώπης όταν καταρρεύσουν τα συστήματα υγείας γιατί μεγαλώνουν οι πιέσεις καλά Ας, αφήστε, αφήστε, να λέμε, δύο ώρες τα λέγαμε τότε, αλλά θα πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία, να είμαστε σοβαροί, τεχνολογία, χρηματοδότηση, νέες μεθόδους σηματοδότησης, πρικοδότησης, ε, επένδυση στην υγεία, στη, στη, στην κοινοτομία και σε ένα σωρό πράγματα και δεν το κάνουμε αυτό. Αν το κάνουμε αυτό, αλλημονό μας. Για την Κίνα. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε μια σειρά προϊόντων από την Κίνα τα οποία δεν είναι εγκεκριμένα. Κρέας, βόλιο, πρόβιο και τα γαλακτοκομικά περνάνε από συστημικές δοκιμές. Σας διαβεβαιώνω. Κάνουμε ό,τι πρέπει να το χαίρουμε τόσο ώστε τα προϊόντα κινδύνου να υπόκεινται εις έλεγχο. Όλα είναι και πιο συχνά. Όποτε τα λέω με τους συναδέλφους τους Κινέζους επιμένω στα ποιοτικά και με χαρά μου διαπιστώνω ότι και αυτοί προς τα εκεί το πάνε. Αλλάζει η κοινωνία τους. Η αυθονία ε, αυξάνεται, ας το πούμε, και, και, και, και, η ζήτηση. Η οικονομία τους προσανατολίζεται προς τα εκεί, προς την οικιακή κατανάλωση και όχι 100% στις εξαγωγές. Οπότε και να και το ζήτημα του τι ζητάει ο καταναλωτής, άρα πάμε στην ποιότητα και άρα στα προαπαιτούμενα για αυτήν την, ε, ε, την, την, την υγεία, την ποιότητα. Άρα το ρεφρέν που ακολουθώ, το σύνθεμα είναι ποιότητα και υγεία στην πηγή για το κάπνισμα, τον καπνό. Τα ήθελα να έχει ήδη γίνει αυτό. Τα ξέρετε, τα είπαμε. Όμως, επίσης, ευθέως σας λέω και παραδέχομαι ότι είναι μέσα σολομός που πάει κόντρα στο ρεύμα, ανεβαίνει το, το ποτάμι. Σας διαβεβαιώ, θα κάνω ό,τι μπορώ, ούτω ώστε να υπάρξει μια ουσιώδης, μεστή πρόταση για να πετύχουμε τους στόχους μας. Να μειωθεί το κάπνισμα, κυρίως στους, στους νέους και κυρίως τις νέες δυστυχώς αυξάνεται λένε τα στατιστικά στοιχεία Επομένως έχω δεσμευθεί σχετικά με αυτό και θα συνεχίσω να κάνω ό,τι μπορώ προς αυτή την κατεύθυνση τώρα όσον αφορά αυτά τα νέα διατροφής τα νέα τρόφιμα όπως προείπαμε να μην επαναλαμβάνουμε τα ίδια ε, περιμένω εσείς τι θα μου πείτε σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα. Θα ήθελα όσο γίνεται συντομότερα κάτι να γίνει. Περιμένουμε. Προτιμώ να περιμένουμε. Πάντως σας λέω, περιμένω τη δική σας απόφαση. Όχι, δεν πρόκειται να διατυπώσω νέα πρόταση. Τώρα για την μη εφαρμοστή σαν νομοθεσία. Έτσι είναι. Το θέμα είναι τι μπαστούνι έχουμε το καρότο. Το μπαστούνι μας το δίνει η νομοθεσία. Και ενίοτε μπορούμε να κάνουμε κάτι. Όμως, όσον αφορά κάποιες μεθόδους, κάποια στοιχεία ελέγχου, ναι, μπορούμε να πιέσουμε πολύ. Όμως, πριν το τέλος της μεταβατικής περίοδου δεν μπορούμε να αναλάβουμε καμία πρωτοβουλία για, τις, την οδηγία για αυτή, για, για τις οτόκες όνειτες. και τώρα... Τίποτα δεν μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος ενός ότος έτους, δηλαδή πριν το τέλος της μεταβατικής περίοδου. Περιμένω να δούμε τι, τι κάνουν τα κράτη-μέλη. Ήδη Ήδη, ήδη το, το, το λέω, οχλώ τα κράτη-μέλη. Να πιέσουν. Και εμείς πιέζουμε τόσο τουλάχιστον να ξέρουμε τι στοιχεία υπάρχουν όσον αφορά την τήρηση της νομοθεσίας. Το σχετικά με το, με, σχέδιο δράσης που έχουμε θα πρέπει να συζητηθεί το τι θα κάνουμε. Και έτσι να, να τι θα κάνουμε και να μην παρακολουθείτε κανένα για αυτά που θα κάνουμε. Επομένω, το πρόβλημά μα θα είναι για το χείριο το πώ θα γίνονται οι έλεγχοι τότε. Και εσείς επομένως πιέστε στις χώρες σας ο καθένας σε σχέση με την εφαρμογή της οδηγίας. Α, αύριο θα πάω στο Λουξεμβούργο, θα μιλήσω με τους υπουργούς Γεωργίας και σας διαβεβαιώ ότι κατηγορηματικά θα τα θέσω όλα αυτά. Και γι' αυτό και για το κρέας αυτό και για όλα τα άλλα που πρέπει να εφαρμοστούν. Αλλά σας είπα. Η εμπειρία μου από τις οτόκες όρνηθες είναι ότι θα πρέπει να προσέξουμε πώς θα νομοθετούμε στο μέλλον. Δηλαδή, όταν βάζουμε 12 ετή μεταβατική περίοδο, εντάξει. Καταρχήν δεν έχω καμία ένσταση κατά αυτού. Όμω προσοχή. Θα πρέπει αυτό να συνοδεύεται από ένα πρόγραμμα δράση. Και με κάποιο χρονοδιάγραμμα παρακολούθηση του γίνεται στα κράτη-μέλη. Και όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, θα πρέπει κάποια αρχή να παρεμβαίνει. Όταν νομοθετούμε, να νομοθετούμε έχοντας υπόψη και το θέμα των ελέγχων. Να εξασφαλίζουμε ότι η νομοθεσία θα εφαρμόζεται στα κράτη-μέλη. Έχετε δίκιο σαν αφορά το πρόγραμμα για περιβάλλον και υγεία. Διότι πρόκειται, όπως είπατε και εσείς, για θέματα πάρα πολύ σχετικά. Η μόλυνση, η ρήπανση, ας πούμε, από, από, τους βόθρους. Όλα, όλα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά για την υγεία. Άρα θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Για το σολάρι, ας πούμε, θεσπίσαμε ένα κανονισμό για να περιορίζεται η ένταση. Η ένταση αυτών των υπεριοδών ακτίνων στην Ευρώπη σε κάθε σολάριο. μάρα και αυτό μας απασχολεί. Evans. Προβλέπεται μια τεχνική λύση ούτως ώστε για τις ζωοτροφές να υπάρχει έλεγχος, μέτρηση, ό,τι χρειάζεται και συλλέγουμε ήδη τα στοιχεία. Ό,τι σχετίζεται με αυτήν την λύση. Πρόκειται ε, να διατυπώσουμε προτάσεις για ανάλογες τέτοιες τεχνικές ε, ε, μεθόδους μέτρησης και για τα τρόφιμα προσδίδει για ανθρώπους. Κυρία Αγίους, όσον αφορά τη μεταφορά των ζώων, το τα έχουμε πει. Και βέβαια λαμβάνει υπόψη την άποψή σας. Uh, ναι, και η ΕΦΣΑ μας έχει παράσχει συμβουλές σχετικά. Αλλά βέβαια έχετε πολλές ερμηνείες η γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Καλό μεταχείριση των ζώων. Είναι θέμα σημαντικό. τώρα κατοχυρώνεται και από τη συνθήκη της Λισαβόνας πρόκειται περί αξίας περί ιδιόδους που είχε ασπαστεί η Ευρώπη έχουμε και την καλομεταχείριση των ανθρώπων βέβαια όπως είπατε το μεν εξαρτάται από το δε αν είναι ναι, καθεν πιστεύουμε πιστεύαμε ότι η καλομεταχείριση των ζώων κατοχυρώνει την ασφάλεια των τροφίμων. Τα έλεγα χθε στην Κοπενχάγη ότι η απονομή αρμοδιοτήτων και εξουσιών είναι, είναι, είναι αυτή η αποκέντρωση ας την πούμε είναι κάτι απαραίτητο γιατί ο κόσμος έχει αλλάξει δεν θέλει να από καθέρα του μιλάμε άρα Μιλάμε για πληροφόρηση. Αλλά όχι μόνο πληροφόρηση. Γιατί θα πρέπει κανείς να ξέρει πώς θα ερμηνεύσει την πληροφόρηση ή να ξέρει πώς εφαρμόζεται στο πρόσωπό του. Και αυτό ισχύει για όλους. Και για την ετικετοθεσία των τροφίμων, για τους ασθενείς. Αυτό επομένως είναι το σημαντικό. το πώς επομένως θα αναβαθμίσουμε, θα ενισχύσουμε το ρόλο του καταναλωτή και του ασθενούς όσον αφορά το τομέα της υγείας επομένως. Και για τη Γεωργία, συνεργάζομαι αρμονικά με τον αρμόδιο συνάδελφο. Τι να πω. Ε, έχει, πολλά να κάνει, δεν μπορώ να, τον, να του φορτώνω κι άλλα αλλά καταλαβαίνω που το πάτε. Ευχαριστώ. Τελευταίο γύρο τώρα Ερωτήσω να τους συναδέλφους. Παύελ Πακ, Κρήτον Αρσένης, Σανούνης Μέρκης. Ε, Mr. Sonic, Mr. Fialna and uh, Madame Okuni, last but not least. Please, Pavel. Thank you, Chair. Pavel, ευχαριστώ. Θέλω να ευχαριστήσω τον Επίτροπο για την Επιτροπή για όλες τις προσπάθειες που καταβάλλετε στην καταπολέμηση του καρκίνου. Πολύ σημαντικό θέμα. Είναι σημαντικό να σκεφτούμε πώς θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα που υπάρχει για τον καρκίνο. Ε, ο διάδοχος θα πρέπει να, έχει, να είναι καλύτερα προσδιορισμένος και πέστε το όπως θέλετε αυτό το πρόγραμμα, το διάδοχο πρόγραμμα. Δεν θα, έχω, δεν θα σας φέρω αντιρρήσεις. Ο Ευχαριστώ, Επίτροπε, που ήρθατε. Ερώτησα τους πολίτες στην Ελλάδα τι να, τους, τι να σας ρωτήσω και μου είπαν διάφορα θέματα. Καταρχάς, η κινητή τηλεφωνία. Έχουμε την έγκαιρη προειδοποίηση. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ομάδες ανθρώπων, όπως οι έγκυες γυναίκες, οι νέοι, στις αρχές 20 και κάτι ας πούμε, ακόμα και οι έφηβοι, που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερους κινδύνους. Το, το hand-free hand -free ή το bluetooth ας πούμε, αυτές οι τεχνολογίες αυξάνουν τον κίνδυνο. Όταν έχουμε καλό σήμα, όταν δεν χρησιμοποιούμε το το τηλέφωνο, μέσα σε αυτοκίνητα τα οποία κινούνται, ε, μέσα σε μεταλλικό περιβάλλον, τότε μειώνεται ο κίνδυνος. Πώς θα ενημερώσουμε τους πολίτες για τον τρόπο μετριασμού των κινδύνων, Γιατί αν δεν ξέρουν, ο κίνδυνος αυξάνεται. Θέλουμε να μας πείτε πώς θα τους ενημερώσουμε. Για τους γάμματα αφόμικρων, οι πολίτε ε, ζητούν υποχρεωτική ετικετοθεσία προϊόντων από ζώα τα οποία τράφηκαν με γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα. Πότε θα κάνει τις προτάσεις Κομισιόν. Τέλος. Ένα σημαντικό θέμα για την Ελλάδα. Τα γενώσιμα φάρμακα. Πολλοί γιατροί λένε δημόσια στην Ελλάδα ότι τα γενώσιμα είναι λιγότερο αποτελεσματικά από αυτά προστατεύονται από διπλώματα ευρεσιτεχνίας, ε, ότι τα γενώσιμα είναι επικίνδυνα. Σχόλιο παρακαλώ. Σανούνι και η λυπη, Ανδρέα Σανώνη. Ευχαριστώ που ήρθατε να απαντήσετε στις ερωτήσεις μας. Θέλω να σας θέσω ένα θέμα που αφορά την διατροφική ασφάλεια των νεογνών. Πρόσφατα εμφανίστηκε διοξίνη στο μετρικό γάλα σε σημαντικές ποσότητες. Ανησύχησαν οι πολίτες και οργανώσεις ε, γιατρών ασχολήθηκαν με αυτό το θέμα. Και μάλιστα έγινε στη Ρώμη και μια διάσκεψη για τη διοξινή στο μητρικό γάλα. Τα παιδιά μας, μόλις γεννιούνται δηλαδή, αρχίζουν να τρέφονται με τρόφιμα τα οποία είναι μολυσμένα με διοξίνη. Ε, υπάρχουν και πιστοποιητικά ανάλυση που το πιστοποιούν. Ε, αυτό προκύπτει ε, σε γυναίκες οι οποίες ζουν ε, δίπλα σε αποτεφρωτές κτλ. Είναι σημαντικό αυτά τα, αυτές οι καταστάσεις να σέβονται τους κανόνες. Επίσης μην ξεχνάτε ότι εκτίθεται ο κόσμος ε, σε ένα κοκτέιλ από μολύνσεις περιβαλλοντικές. Θέλω να σας ζητήσω να μου πείτε αν γνωρίζετε αυτή την κατάσταση και αν τη γνωρίζετε τι πιστεύετε για αυτό το πρόβλημα. Τι μπορείτε να κάνετε ούτω ώστε να επιλύσετε αυτό το ζήτημα το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γκράτσια, γερμανιστή. Επόμενο ομιλητή. Ευχαριστώ που ήρθατε. Ε, μια στιγμή πρώτη κυρία, η Γιούντιτ. Μέρκες. Γιούντιτ, ευχαριστώ Επίτροπε που ήρθατε και που μας απαντήσετε σε αυτό το βομβαρδισμό ερωτήσεων με τις οποίες σας πυροβολήσαμε. Έχω και, άλλους, και άλλες ερωτήσεις. Πρώτον, τα νανοσωματίδια και την νανοτεχνολογία. Δεν έχουμε μια συγκεκριμένη στρατηγική Δεν υπάρχει δικό χάρτη του 2015 για τα νανοσωματίδια. Είναι και ώρα να αποκτήσουμε. Γιατί το νάνο θα το βρούμε μπροστά μα. Είναι θέμα του μέλλοντο. Και όλε οι πτυχέ τη νανοτεχνολογία που δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα θα μα απασχολήσουν. Ε, διαλύονται τα νανοσωματίδια, παράδειγμα χάρη του αργύρου, στο περιβάλλον. Και κλείονται στο περιβάλλον. Με συνέπειε που δεν έχουν μελετηθεί 100%. Είδαμε ήδη ότι ο Άργυρος μειώνει την ε, γονιμότητα κάποιων ζώων. Και νομίζω ότι τα νοσοματίδια πρέπει να τα προσέξουν περισσότερο, όχι μόνο για την υγεία των ανθρώπων, αλλά και των ζώων. Ζητώ λοιπόν να υπάρξει νομοθεσία, τουλάχιστον κανονισμός. Ο κύριος Ταγιάννη είναι υπεύθυνο ε, για το θέμα αυτό. Αλλά μια και συνδέεται πολύ με την υγεία αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να το θέσω και σε εσά και να μου πείτε, θα υπάρξει κανονισμό για την αντιμετώπιση του θέματος αυτού και την ετικετοθεσία. Επίσης, για τις ζωοτροφές και το σανό. Μπορούμε να αλλάξουμε το σανό που τρώνε τα ζώα ούτω ώστε να συνεισφέρουμε σε λιγότερη έκκληση δίωξη του άνθρακα. Τέλο. στην ακρόαση, την πρώτη φορά που ήρθατε στο Κοινοβούλιο, σα μίλησα για την μεταφορά των ζώων. Θέλω να επανέλθω τώρα σε αυτό. Τότε μου είχατε απαντήσει στην ακρόαση ε, μου είχατε πει εκείνη τη χρονιά ότι μέχρι το τέλος εκείνης της χρονιάς θα υπάρχει νομοθεσία. Αυτό έγινε το 2010. Πούντι, Σόνικ. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ για την οδηγία του καπνού που αναφέρατε κύριε Πρόεδρε και είπατε πως ε, κάτι έπρεπε να γίνει για να μειωθεί η ελκυστικότητα των τσιγάρων ε, θα μπορούσαν ακόμα και να απαγορηθούν ε, αν είναι γλυκά ας πούμε ή αρωματισμένα ή περιέχουν εθιστικές ουσίες Υπάρχουν όμως ουσίες οι οποίες ε, ε, χρησιμοποιούνται και χρησιμοποιούνται στην διαδικασία αυτή και αναρωτιέμαι αν τις έχει λάβει υπόψη η Κομισιόν. Τα τσιγάρα με γεύση μέντα, παραδείγματο χάρη, υπάρχουν στην Πολωνία εδώ και 100 ε, χρόνια περίπου και στη Φιλανδία. Δεν νομίζετε λοιπόν πως η παράνομη παραγωγή αυτών των τσιγάρων θα μπορούσε να προκαλέσει πρόβλημα. Ευχαριστώ. Χέλνερ. ευχαριστώ. Θα αναφερθώ και εγώ στα προϊόντα καπνού. Τα έχουμε συζητήσει για το άρθρο 8 και την απαγόρευση του καπνού που μασάνε στη Σουηδία. Παρά το ότι βλάπτει λιγότερο από το ε, τσιγάρο. Αναρωτιέμαι τι, αν, τι θα έλεγαν οι Γάλλοι αν απαγορεύαμε το κόκκινο κρασί και του λέγαμε ότι η βότκα δεν πειράζει. Τέλο πάντων, την προηγούμενη εβδομάδα τα σουηδικά ΜΜΕ είπαν πως ε, θα απαγορευτούν αρωματικές ουσίες που είναι απαραίτητες για το σνούς, τον καπνό αυτό που έχουμε στη Σουηδία και μάλιστα παρακάμπτεται η, η συνθήκη ένταξης της Σουηδίας γιατί είχε προβλέψει ρητά αυτό το προϊόν, αλλά δεν απαγορεύεται το προϊόν, αλλά αυτά τα οποία χρειάζονται για να φτιαχτεί. Μα ένα εκατομμύριο από τα 9 εκατομμύρια Σουηδού το χρησιμοποιούν και του λέτε πρέπει να το κόψετε. Ε, δε. Ναι. Εντάξει, μπορεί να πρέπει, αλλά όχι να του αναγκάσει η Κομισιόν. Οπότε, μπορείτε να ξεκαθαρίσετε, να υποσχεθείτε πως αντί ε, να συζητήσουμε την απαγόρευση του σνούς από την πίσω πόρτα θα μπορούσαμε να μεταχειριστούμε όλα τα προϊόντα καπνού με τον ίδιο τρόπο τουλάχιστον. Ευχαριστώ. Η κυρία Οκονή τελευταία. Merci, Président, Monsieur le Commissaire. Ευχαριστώ, Επίτροπε. Όλα τα θέματα που ήθελα να θίξω παρουσιάστηκαν ήδη από άλλους. Ήθελα να μιλήσω για τον καπνό, ήθελα να μιλήσω για τα εισαγόμενα από την Κίνα. Ήθελα να μιλήσω επίσης για τις οτόκες όρνηθες. Όλα τα συζήτησαν οι συνάδελφοι. Κύριε Πρόεδρε, με ακούτε. Θα ήθελα τότε να μου υποσχεθείτε ότι την επόμενη φορά θα είμαι η πρώτη που θα πάρει το λόγο για να ρωτήσω τον Επίτροπο. Γι αυτό με αυτόν τον τρόπο ε, θα είμαι σίγουρη ότι θα μιλήσω. Τώρα αφήνω την θέση μου σε έναν άλλο συνάδελφο. Ναι. Ε, την άλλη φορά, για εκεί που κάθεστε την άλλη φορά μόλις σηκώσετε το χέρι θα σας δω πρώτη. Λοιπόν κύριε Επίτροπε, σας παρακαλώ, α, περιμένουμε τις απαντήσεις σας. I, uh, I gladly come here. Με χαρά έρχομαι εδώ για να σας εξηγήσω τι κάνουμε. Να απαντήσω σε ερωτήσεις και είμαι στη διάθεσή σας να μου στέλνετε σχόλια και στο μεταξύ, έτσι. Δεν σπάει ο διάλογος μόλις φύγω από εδώ. Είμαι ανοιχτό. Θέλω να ακούσω ιδέες από εσά και ερωτήσεις. Και να προσπαθήσω να κάνω διάλογο. Ούτως ώστε να εμπλουτίσω και το δικό μας προβληματισμό γιατί νομίζω ότι είναι και για τι μελλοντικέ μας πολιτικές. Δηλαδή, συνεχή επαφή με εσά, συνεχή ερωτήσεις. Μην περιμένετε, λοιπόν, να σα δώσουν το μικρόφωνο. Όποτε θέλετε, ελάτε σε επαφή μαζί, μαζί μου, γιατί είμαι στη διάθεσή σας. Κύριε Πάβελ, κάνετε κάποια σχόλια για τον καρκίνο και άλλα πράγματα. Ο κύριος Ασένης έκανε κάποιες ερωτήσεις για τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία. Να σας πω ότι αυτά τα θέματα είναι αρμοδιότητα του κράτους μέλους. Ο τρόπος που θα διαχειριστεί αυτά τα θέματα, η πληροφόρηση που θα δώσει για το μετριασμό του κινδύνου είναι θέμα του κράτους μέλους. Αλλά καταγράφω αυτό που είπατε και αυτή τη στιγμή Ζητάμε από την Επιστημονική μας Επιτροπή να αναθεωρήσει όλο το θέμα των ηλεκτρομαγνητικών πεδίων. Και είμαι σίγουρος ότι ανάλογα με το τι θα μας πει η Επιστημονική Επιτροπή, θα δράσουμε προς το συμφέρον των πολιτών. Και θα τους ενημερώσουμε για το πώς μπορούν να μειώσουν όσο μπορούν περισσότερο οποιονδήποτε κίνδυνο από τα κινητά τηλέφωνα γιατί τα κινητά τηλέφωνα είναι παντού σήμερα. Τα χρησιμοποιούμε παντού. Ακόμα και εξάχρονα έχουν κινητά. Γεννιούνται με τα κινητά. Είναι, δεν είναι σχεδόν ε, θέμα επιλογή των γονιών, έχει ξεφύγει τα χέρια τους. Το θέμα είναι να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους για το πώ θα τα χρησιμοποιούν, όπως ε, εκπαιδεύουμε ανθρώπου για να χρησιμοποιούν άλλα εργαλεία. Για την επισήμανση των γάμα ταφόμικρων, η υποχρεωτική ετικετοθεσία των γάμα ταφόμικρων και προϊόντων όπως το γάλα και το κρέας ή ζώων που έχουν ε, τραφεί με τρόφιμα γάμα ταφόμικρων, ο κίνδυνος δεν έχει επιστημονική βάση. φαίνεται ότι η ζωοτροφή που προέρχεται από τέτοια ζώα δεν ξεχωρίζει τις ζωοτροφές ε, τις υπόλοιπες. Ένα ζώο που το θρέψαμε με γάμα όμικρον και ένα ζώο που το θρέψαμε με μη γάμα όμικρον, όταν αναλύσουμε τα προϊόντα που παράγουν, δεν υπάρχουν καθόλου διαφορές. Δεν προβλέπεται. Οπότε θα αξιολογήσουμε και θα μελετήσουμε τις πρωτοβουλίες που υπάρχουν τώρα για τους οργανισμούς αυτούς και θα προχωρήσουμε προς περαιτέρω εναρμόνιση φέτος γιατί επίσης προσπαθούμε να δούμε μέχρι πού μπορούμε να φτάσουμε σε αυτό το μέτωπο τώρα όσον αφορά τις διοξίνες στις παιδικές τροφές. Έχουμε όσο γίνεται πιο αυστηρές διατάξεις σε όλο τον κόσμο. Και καθόμαστε και παρακολουθούμε προγράμματα τα οποία εντοπίζουν την επιμόλυνση από τις διοξίνες. Και αν επισημαθεί ένα τέτοιο προϊόν, αποσύρεται. Υπάρχει επομένως υποχρέωση δοκιμής για διοξίνη και άλλες ουσίες. Α, Φερρυπίν, πέρσι έγινε αυτό στη Γερμανία. αν επισημανθούν, κινητοποιεί το σύστημα το οποίο όσον αφορά την ανείχνευση λειτουργεί ανοιχνεύουμε, εντοπίζουμε και αποσύρουμε. Υπάρχει στο περιβάλλον και πολλές φορές συμβαίνουν τέτοια μόλις, μόλις. Όμως εμείς, εμείς επαγρυπνούμε διαρκώς. Υπάρχει έλεγχος ολοκληρωτικός παντού. Νανοτεχνολογία. Και επ' αυτού βέβαια... Είμαι συναρμόδιος. Πρέπει να δούμε τα θέματα νανοτεχνολογίας. Πρέπει να το ξαναπώ. Η οδηγία για τα νέα τρόφιμα, για τα novel food, την οποία ανέφερα. Έχω, έχει το πρώτο βήμα για την καταπολέμηση της νανοτεχνολογίας. Αυτή τη μάχη μου τη χάσαμε, γιατί δεν συμφωνήσαμε. Και αυτό, για αυτό το λόγο πιέζω τόσο ώστε αυτή η οδηγία να προχωρήσουν να δουν πιο γρήγορα. Χωρίς να περιμένουμε. Υπάρχουν πολλά στοιχεία που είναι χρήσιμα για τους καταναλωτές. Και είναι κρίμα που την αφήνουμε αυτή την ε, νομοθεσία στο λίμπο. Ασχολούμαστε με άλλα πράγματα, κλωνοποίηση και Τέλο πάντων, δικό σα θέμα. Εσεί αποφασίζετε, όχι εγώ. On, ε, and on transport. Για την ε, νομοθεσία για τις μεταφορές. Σε τι δεσμευτήκαμε. Να εκδώσουμε μία έκθεση για τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζονται οι σχετικοί κανονισμοί. Το κάναμε. Και όπως είπα προηγουμένως, πρέπει να βρούμε τη σωστή λύση για τη μεταφορά των ζώων. Για μένα, πρέπει να θέσουμε σε συζήτηση το ζήτημα της μεταφοράς. Γιατί η μεταφορά και για το σανό των ζώων θα πρέπει να το δούμε. Κύριε Σόνι, καπνός. Ε, διαφοροποιούμε ανάμεσα σε χαρακτηριστικές γεύσεις, βανίλια, σοκολάτα, πινακολάντα, ε, διάφορες αρωματικές ουσίες. Τις διακρίνουμε αυτές. Το διαφοροποιούμε αυτό και άλλα συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα στην παραγωγή αυτού του καπνού. Ξέρουμε ότι κάποια είδη καπνού θα πρέπει να αναβαθμιστούν με τη χρήση κάποιων ουσιών. We are making the difference in that regard. Um, Επομένως κάνουμε τη διάκριση. Ναι. Και φυσικά το μεντόλ, η μέντα, είναι κάτι που συζητήσαμε, όπως και οι άλλες αρωματικές ουσίες. Και τώρα πρέπει να πάω στο παράνομο τμήμα αυτής της ερώτησης, στο παράνομο, την παράνομη διάσταση. Προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε την ιχνηλασιμότητα των προϊόντων καπνού, ούτως ώστε να καταπολεμήσουμε το λαθρεμπόριο καπνού και το, τις απομιμήσεις και το λαθρεμπόριο. Και δεν το κάνουμε για φορολογικούς λόγους, γιατί δεν θέλουμε φθηνοτσιγάρες αγορές μας. Υπάρχει θέμα πρόσβασης που και εκεί προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε. Το, ο σουηδικός καπνός σνούς είναι ένα μόνιμο ζήτημα. Η πραγματικότητα είναι αυτή. Υπάρχει απόφαση του δικαστηρίου για αυτό το σνους. Αυτό ισχύει, αλλά υπάρχει παρέκκληση για το σουηδικό σνους και δεν πρόκειται να φύγει ούτε από την μπροστινή πόρτα ούτε από την πίσω. Αν θέλετε όμως να βάλετε γεύση σοκολάτα στο σνούς, ε, αυτό θα το απαγορεύσουμε, γιατί προσπαθούμε να το απαγορεύσουμε και στα τσιγάρα. Ευχαριστώ πολύ, Επίτροπε, για τις απαντήσεις σας. And for the possibility to have an exchange για τη δυνατότητα αυτή που μας δώσατε να ανταλλάξουμε απόψεις. Εμείς ασχολούμαστε και με το περιβάλλον και με τη δημόσια υγεία και με την ασφάλεια των τροφίμων. Ο Τζο Λάινεν ήταν ε, ε, υπεύθυνο για την έκθεση πρωτοβουλίας για αυτά τα θέματα. Πρέπει να ξεκινήσουμε το περιβάλλον και μετά να πάμε στην υγεία. Γιατί αυτά τα θέματα είναι αλληλένδετα. Και για την ασφάλεια των ε, τροφίμων και όλα τα άλλα θέματα, τον καπνό, θα έχουμε σκληρές συζητήσεις. Είσαστε υπεύθυνο για την πολιτική υγεία. Είσαστε υπεύθυνο και για την πολιτική καταναλωτών. Αυτές οι πολιτικέ που αφορούν 500 εκατομμύρια πολίτες. Θέλουμε να τους δείξουμε ότι βελτιώνουμε και τα πρότυπα υγείας και τα περιβαλλοντικά πρότυπα και τα πρότυπα για τα τρόφιμα.